Καλημέρα σας. Καλημέρα σε αγαπητοί συνάδελφοι. Ο πρόεδρος μου ζήτησε να προεδρεύσω εγώ διότι ε, έχει κάποιες σημαντικές συνειδημένες υποχρεώσεις. Ας με λοιπόν για το υπόλοιπο της ε, συνεδρίασης. Έχω βέβαια τις ηγετικές ικανότητες ε, του κυρίου Μπούζεκ. Ο συνήθως, ο κύριος Μπούζεκ κάνει μια δοκιμαστική ψηφοφορία, επομένω θα κάνω και εγώ το ίδιο. Ας α, ψηφίσουμε λοιπόν δοκιμαστικά. Χρησιμοποιήστε παρακαλώ πολύ τις κάρτες σας. Και να η ερώτηση επί της οποίας μπορείτε να αποφανθείτε. Πιστεύετε ότι ο πρόεδρος Τραμπ έχει κάνει μια καταπληκτική δουλειά κατά τη διάρκεια των πρώτων εβδομάδων ε, της θητείας του. Μπορείτε να ψηφίσετε από αυτού του ερωτήματος. Άρτη ψηφοφορία. Πέρας. 11. Η επόμενη ερώτηση, ποιος ψήφισε έτσι. Λοιπόν, πολύ ωραία. Ας προχωρήσουμε στις ψηφοφορίες. Πρώτη έκθεση, η έκθεση της κυρίας Κομπούλα Νάτρη σχετικά με τους κανόνες που διέπουν τις αγορές περιαγωγής χονδρικής. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Άρτη ψηφοφορία. Πέρας. Όχι ακόμα. And did you vote in favor? Yes? Okay. Ψηφίσατε υπέρ. Πέρας. υπέρ, ένας κατά τρεις αποχές, συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια κυρία Κουμπούλα Νάτρη. Περνάμε τώρα στη δεύτερη ψηφοφορία που έχει να κάνει με το σχέδιο δράσης Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Η συγγήτρια είναι η κυρία Αγγέλικα Μιλινάρ, άρτη ψηφοφορία, αψηφίζουμε κανονικά. Συμβαστική τροπολογία παριθμών 1, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική παριθμών 2 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 13 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική υπερθμών 3 υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 17 υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία υπαριθμών 4 υπέρ παρακαλώ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 5 κατά, υπέρ, με συγχωρείτε, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική υπερθμόν 6 υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 7 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 46 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 47 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 48 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 49 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 59 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 61 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 63 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 9 υπέρ παρακαλώ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 67. Έχουμε εδώ πέρα προφορική τροπολογία. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 73 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 74 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά παρακαλώ. Άρτη ψηφοφορία. Πέρας. 43 υπέρ, μία ψήφος κατά και έξι αποχές. Συγχαρητήρια στην εισηγήτρια. Ολοκληρώνονται εδώ πέρα ψηφοφορίες. <clears throat> Okay, now I get to the... Πολύ ωραία. Point number 10. Σημείο 10 ενεργειακή απόδοση των κτηρίων. Να σας ενημερώσω ότι στις 30 Νοεμβρίου η Κομισιόν παρουσίασε τη δέσμη για την καθαρή ενέργεια για όλους τους Ευρωπαίους συμπεριλαμβανομένων οκτώ νομοθετικών προτάσεων που καλύπτουν ενεργειακή απόδοση, ανανεώσιμες ενέργειες, το σχεδιασμό αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, ασφάλεια εφοδιασμού ηλεκτρικής ενέργειας και κανόνες διακυβέρνηση για την Ενεργειακή Ένωση. Στη σημερινή συνάντηση θα αρχίσουμε τη δουλειά της Ήτρε πάνω σε αυτό το νομοθετικό πακέτο, συζητώντας δύο από τις προτάσεις. Θα αρχίσουμε με μια ανταλλαγή απόψεων επί της προτάσεως αναθεωρημένης οδηγίας ε, για την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων, έκθεση Μπένσεν. Μετά θα κάνουμε μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων πάνω στην πρόταση οδηγίας για την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Αυτή είναι η έκθεση Μπλάνκο Λόπες. Και οι άλλες προτάσεις της δέσμης θα συζητηθούν στην Επιτροπή στις συνεδριάσεις μας τον Μάρτιο και τον Απρίλιο. Προβλέπεται μία ώρα συζήτηση τώρα για αυτό το θέμα και δίνω το λόγο στον κύριο Μπέντσεν, ο οποίος θα παρουσιάσει τις πρώτες απόψεις του ε, για την πρόταση αναθεωρημένης οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων. Έχετε πέντε λεπτά κύριε Μπένσεν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ την Επιτροπή για την εξαιρετική πρόταση σχετικά με την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων. Νομίζω ότι ακόμα διαμορφώνουμε απόψεις ε, και θα ακούσω τις προτεραιότητες και των σκιωδών με μεγάλο ενδιαφέρον. Οι βασικές φιλοδοξίες είναι σαφείς όσο πιο αποδοτικά τα κτίρια, τόσο μικρότεροι λογαριασμοί ηλεκτρικής ενέργειας, θα μειωθεί η κατανάλωση, θα, μειωθούν, θα μειωθούν οι εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα, θα είμαστε λιγότερο εξαρτημένοι από εισαγωγές. Σήμερα οι εισαγωγές στοιχίζουν ακριβά, ιδιαίτερα εισαγωγές από τον κύριο Πούτιν. Οι, θα μειω, μειωμένοι λογαριασμοί θα μειώσουν και την εξάρτηση και θα αυξήσουν την πολιτική μας ασφάλεια. Οι ανακαινήσεις μπορούν επίσης να δημιουργήσουν απασχόληση ε, ιδιαίτερα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ας τα βάλουμε σωστά τα πράγματα. Εστιάζομαι σε τρία σημεία που πιστεύω ότι πρέπει να τα δούμε πολύ προσεκτικά. Το πρώτο είναι ο μακροπρόθεσμος σχεδιασμός, δεύτερον ε, εξασφάλιση χρηματοδότησης και τρίτον ε, μελλοντικές αποφάσεις. Μακροπρόθεσμος σχεδιασμός. Εδώ χρειάζεται στρατηγική, θα πρέπει να επιτύχουμε τους κλιματικούς στόχους για το 2050. Γι' αυτό τα κτίρια πρέπει να συμβάλλουν περισσότερο. Η Κομισιόν λοιπόν με βρίσκει απόλυτα σύμφωνο όταν θέλει να υποχρεώσει τα κράτη-μέλη να καταρτήσουν στρατηγικές ανακαίνησης των κτηρίων στα πλαίσια των σχεδίων για την ε, πολιτική ενέργειας. Θα πρέπει επίσης να δεσμευτούν τα κράτη-μέλη και να έχουν ε, αποτελέσματα στα πλαίσια της επικουρικότητας βέβαια. Θα πρέπει να ε, στηριχθούμε ε, με τρόπο αποτελεσματικό από άποψη κόστου στα υφιστάμενα κτίρια. Θα πρέπει να δείξουμε κατανόηση βέβαια στο κόστος που πρέπει να καταβληθεί. Από την άλλη η ανακαίνιση των κτιρίων είναι πολύ σημαντική. Ε, στην ε, χώρα μου οι φόροι είναι πάρα πολύ υψηλοί, ε, όχι τόσο η συμβολή στην ενεργειακή απόδοση. Εδώ υπάρχει μεγάλο περιθώριο πολλές φορές, δηλαδή τα θέματα πρέπει να τα δούμε σε εθνικό επίπεδο. Για τη χρηματοδότηση είμαι ευγνώμων, διότι η Κομισιόν έχει τη φιλοδοξία να αρχίσει επενδύσεις στις ανακαινήσεις κτηρίων. Οι υποχρεώσεις των κρατών μελών ε, είναι να δημιουργήσουν μακροπρόθεσμες στρατηγικές και ένα κατάλληλο πλαίσιο. Πολύ λογικές προτάσεις. Θεωρώ ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε με σωστές βάσεις στην αναθεώρηση της οδηγίας. Ε, σημαντικό είναι το θέμα της ιδιωτικής χρηματοδότησης. Θα πρέπει οπωσδήποτε να είναι αποτελεσματικές ιδιωτικές επενδύσεις και αυτό θα γίνει ενεργοποιώντας ορισμένα ε, συνταξιδοτικά ταμεία, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και για να ε, λειτουργήσουν οι πόροι θα πρέπει να υπάρχει σαφής προδιαγραφή για τη χρήση. Ε, θα πρέπει να τεκμηριώνεται επίσης ε, το αποτέλεσμα της ανακαίνησης συγκρίνοντας πριν και μετά την κατάσταση και τα πιστοποιητικά. Ε, χρειάζεται ενεργειακό πιστοποιητικό μετά την ανακαίνιση αλλά πρέπει να παρακολουθούμε και τις μικρότερες ανακαινήσεις. Ας πάμε στο τρίτο σημείο σχετικά με τις μελλοντικέ αποφάσεις. Όλοι συμφωνούμε ότι θα πρέπει να ε, υπάρχουν και άλλα μέτρα πέρα από τη μείωση του, ε, της χρήσης του άνθρακα. Χρειάζεται λοιπόν κατάλληλη υποδομή. Ε, πρέπει να διασφαλίσουμε ε, με μελλοντικές οδηγίες τη σωστή λειτουργία και τη χρήση της νέας τεχνολογίας. Ε, είναι σημαντικό επίσης να συμπεριλάβουμε τη χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας στα κτίρια. Αυτό θα βοηθήσει και τις επιθεωρήσεις και θα υπάρχει περισσότερο ε, ευφυής χρήση των τεχνολογιών. Προσβλέπω στη συνεργασία με τους Σκιώδης, ε, θέλω να ακούσω όλες τις απόψεις σας ε, σχετικά με την πρόταση της Κομισιόν, σχετικά με τις προτεραιότητες που τίθενται και πώς ε, αντιμετωπίζουμε τη δυναμική που ανοίγεται σε αυτό το τομέα. Να μειώσουμε τους λογαριασμούς, να κάνουμε άλματα στην ενεργειακή απόδοση, να επιτύχουμε τους στόχους ε, στον τομέα της ενέργειας για μια ε, πιο ανεξάρτητη και ασφαλή Ευρώπη. Ευχαριστώ, ευχαριστώ που τηρήσατε και το χρονικό όριο. Τώρα, η κυρία Κομπούλα Νάτρη από τους Σοσιαλιστές. Δύο λεπτά. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, θα μιλήσω στη γλώσσα μου τα φιλανδικά αυτή τη φορά. Όπως είπε και ο εισηγητής, είναι θετικός ο αντίκτυπος στην οικονομική ανάπτυξη και στο ισοζύγιο πληρωμών όταν καταβάλλονται προσπάθειες για ενεργειακή απόδοση. Θα βοηθήσουμε και στην ανταγωνιστικότητα και την απασχόληση στον τομέα των κατασκευών. Αυξάνονται επίσης ε, και οι δεξιότητες στον τομέα της κατασκευής έξυπνων κτηρίων. Θα πρέπει να δούμε πώς θα είναι οικονομικά βιώσιμα τα κτίρια όταν ανακαινίζονται. Ένα κτίριο με καλύτερη ενεργειακή απόδοση είναι και πιο ευχάριστο για τους ε, ανθρώπους που το χρησιμοποιούν. Ε, στη Βαρκελόνη ε, ε, χθες τελείωσε ένα συνέδριο σχετικά με την ενεργειακή απόδοση και τα έξυπνα σπίτια. Είναι μεγάλη ευκαιρία αυτή που ανοίγεται για ε, πολλούς τομείς. Ε, δεν μιλάμε μόνο για τείχους, αλλά γενικότερα ενεργειακή διαχείριση και έξυπνα σπίτια. Ε, χαιρετίζω τις ε, ιδέες που μας παρουσίασε ο εισηγητής, με βρίσκουν σύμφωνοι. Εξ ονόματος της ομάδας μου πρέπει να πω ότι είναι σημαντικό να εστιάσουμε και στην ενεργειακή φτώχεια και να εξετάσουμε διάφορα χρηματοδοτικά μοντέλα για τις διάφορες χώρες που θα πρέπει να συμπεριληφθούν στις εθνικές εκθέσεις. Πώς δηλαδή οι χώρες μπορούν να διαχειριστούν και να βελτιώσουν την ενεργειακή φτώχεια. Γιατί υπάρχουν διαφορές σε εθνικό επίπεδο, στα εθνικά συστήματα στήριξης, ε, η χρηματοδότηση ε, εύκολα δηλαδή μπορεί να πάει σε νέα κτίρια ε, που είναι για τους πλούσιους και δεν πάνε σε ενοικιαζόμενα σπίτια όπου ζουν οι πιο φτωχοί. Πρέπει να δούμε όλα αυτά τα μοντέλα χρηματοδότησης όταν κάνουμε ανακαίνιση ε, κτηρίων και σπιτιών που ενοικιάζονται. Ε, συμφωνώ και με το σημείο που αφορά την ε, ηλεκτρονική κινητικότητα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, που μου δώσατε το λόγο συμφωνούμε 100% ότι υπάρχει τεράστιο δυναμικό αναξιοποιείται όταν πρόκειται για την ενεργειακή απόδοση. Το 40% της ενεργειακής απόδοσης ε, αφορά στα κτίρια και πρέπει να συνεχίσουμε να προσπαθούμε να μειώνουμε την κατανάλωση ενέργειας. Εδώ έχουμε μια άλλη πρόταση που αλλάζει τους κανονισμούς σε αυτό το τομέα. Η σύσταση είναι να αναβαθμιστούν τα κτίρια. Υπάρχουν πολλές προσεγγίσεις που προτείνονται στο έγγραφο. Οι λύσεις θα πρέπει να βοηθήσουν στα πλαίσια μακροπρόθεσμου σχεδιασμού να βελτιωθεί η ενεργειακή απόδοση. Οι διατάξεις ε, αφορούν τη χρήση αυτοματοποιημένων συστημάτων και έξυπνων συστημάτων στα κτίρια. Η, η ηλεκτρονική κινητικότητα θα πρέπει επίσης να προωθηθεί με κίνητρα στα συμπατικά κυρίως κτίρια. Αυτά τα λέει το κείμενο. Εγώ θεωρώ σημαντικό να προωθήσουμε την ενεργειακή απόδοση, αλλά δεν αρκεί μόνο αυτό. Θα πρέπει να εξορθολογήσουμε και να απλοποιήσουμε τις θέσεις μας. Καμιά φορά χρειάζεται και η απελευθέρωση, γιατί αυτά που είχαμε μέχρι τώρα δεν έδωσαν ε, καλά αποτελέσματα σε ό,τι αφορά τον έλεγχο, για παράδειγμα, των λεβίτων θέρμανσης. Εκεί δεν λειτουργήσε το σύστημα. Ένα παράδειγμα. Θέλω να πλουστευτούν οι διατάξεις, αλλά οι διατάξεις που αφορούν την ηλεκτροκινητικότητα δημιουργούν κάποιες ανησυχίες. Σε κτίρια που δεν είναι κατοικίες, ένα στα δέκα πρέπει να γίνουν αναπροσαρμογές προς τις απαιτήσει της ηλεκτρονικής κινητικότητας. Αυτό αφορά όλα τα σπίτια που δεν είναι κατοικίες ε, είναι πολύ αυστηρή αυτή η προδιαγραφή. Θα έλεγα ότι αυτή η πρόταση είναι πολύ δαπανήρη. Εμείς θέλουμε να είμαστε αποδοτικοί προπάντων. Η αρχή αυτή θα πρέπει να αφορά και κατοικίες και κτίρια που δεν είναι κατοικίες. Δεν είμαι κατά του εγγράφου καθ' αυτού, αλλά πιστεύω ότι πρέπει να δημιουργηθεί υποδομή με τρόπο ορθολογικό. Και στη διαδικασία αυτή πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και τον κορεσμό στην αγορά. Η ηλεκτρονική κινητικότητα ναι, αλλά πρέπει να δούμε τις ιδιαιτερότητες και τους, τις ε, προϋποθέσεις που ισχύουν στα κράτη-μέλη. Ε, δύο λεπτά, μην τα εξεπερνάτε από την Άλντε. Ευχαριστώ. Να ευχαριστήσω πρώτα τον εισηγητή που ζήτησε και τη γνώμη των σκιωδών από τώρα. Ε, υπάρχουν διάφορες ε, προτάσεις, όπως ήδη τονίστηκε η πρόσβαση στη χρηματοδότηση για την ε, ανανέωση είναι σημαντικό θέμα, αλλά υπάρχουν και άλλα προβλήματα που εμποδίζουν τις καινοτομίες. Πρέπει να καταργηθούν τα διοικητικά εμπόδια που δημιουργούν αντικίνητρα στην ναι, καινοτομία και στην ανανέωση και για τους ιδιώτες αλλά και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις κυρίως. Θα πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι εκεί που υπάρχει χρηματοδότηση είναι και ε, προσιτή. Γιατί κράτη-μέλη, πολλά κράτη-μέλη έχουν πολύ κατακαιρματισμένα συστήματα που μάλιστα διαφέρουν από Δήμο σε Δήμο. Πράγμα που οδηγεί σε κακή ενημέρωση για το, για το είδος των ε, έργων που είναι και εδώ θα πρέπει ε, να μιλήσουμε και για τη δημιουργία των μοναδικών θηρίδων ε, ε, επαφής και ενημέρωσης ώστε να είναι πιο αποτελεσματική η πρόσβαση. Υπάρχουν καλά παραδείγματα και θα πρέπει σε αυτά να βασιστούμε. Επίσης πιστεύω πρέπει να δούμε τον τρόπο με τον οποίο εκτιμούμε τα, τα διάφορα έργα στα πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης. Ε, καθώς επίσης και για τα άλλα θέματα που σχετίζονται με την ενέργεια που λαμβάνουμε, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τα ενεργειακά συστήματα στο σύνολό τους, τα πιο οι πιο αποτελεσματικές ε, λύσεις και από την άποψη του κόστους είναι αυτές που ε, ακολουθούν μια γενική και καθολική προσέγγιση όπου λαμβάνονται υπόψη και τα κτίρια, γιατί τα κτίρια δεν είναι μόνο το περίβλημα, αλλά είναι ε, για μια ε, επιχείρηση, αλλά ε, υπάρχουν δυνατότητες ανανέωσης και στα κτίρια που ήδη είναι κατασκευασμένα και άρα τεράστιες επιχειρηματικές ευκαιρίες αλλά και ευκαιρίες απασχόλησης. Θα πρέπει να είμαστε λοιπόν μέσα, στο, <coughs> μέσα στην Ενεργειακή Ένωση να δημιουργηθούν όλες αυτές οι ευκαιρίες. Προσβλέπω συνεργασία μεταξύ μας. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα ο κύριος που αντικαθιστά τον κύριο Μαρσέλης. Α, όχι. Ο κύριος Μαρσέλης αντικαθιστά τον κύριο Τούρμες ανάποδα. Ναι. Εγώ είμαι ο κύριος Μαρσέλης ε, και θα... Ε, μόλις έφτασα από άλλη επιτροπή για μας, τους πράσινους, ε, έχουμε κάποια βασικά αιτήματα που θα συνεχίσουμε να τα υπερασπίζουμε ε, και βασικά θεωρούμε ότι πρέπει να δούμε πολύ προσεκτικά πώς θα εφαρμοστεί η Συμφωνία του Παρισιού και οι δύο βαθμοί να μην γίνουν ενάμιση ε, ε, με περισσότερες φιλοδοξίες δηλαδή να προσπαθήσουμε να κάνουμε την ε, πραγματικότητα τους στόχους αυτούς που βασίζονται στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας οι στόχοι αυτοί. Αυτός είναι ο βασικός στόχος αυτή τη μεταρρύθμιση. Επίσης, το να σκεφτόμαστε ε, ένα κτίριο ποτέ δεν πρέπει να το βλέπουμε απομονωμένα. Θα πρέπει να το σκεφτούμε μέσα στο οικοσύστημά του το κάθε κτίριο, ότι δηλαδή αυτό συνδέεται με το υπόλοιπο αστικό ε, ε, ή αγροτικό περιβάλλον. Θα πρέπει να είναι δηλαδή διασυνδεδεμένο με το υπόλοιπο σύστημα εντός το οποίο βρίσκεται. Τρίτο, θα πρέπει να θυμίσουμε ότι δεν λύνονται όλα με την τεχνολογία. Η τεχνολογία μπορεί να βοηθήσει απέναντι στην οικολογική και κοινωνική κρίση, αλλά ε, υπάρχουν και του άλλου είδους τεχνολογίες, εκτός από το high-tech και το ε, o-tech, δηλαδή other type of technologies, άλλου είδους τεχνολογίες πιο απλές, πιο προσιτές. Και η τεχνολογία μπορεί να έχει και αυτή οικολογικό αντίκτυπο και πρέπει όλα αυτά να τα λαμβάνουμε υπόψη ώστε να φτιάξουμε μια μεταρρύθμιση γενική λαμβάνοντας υπόψη τον κύκλο ζωής των τεχνολογιών. Επίσης, μιλάμε για επενδύσεις και εδώ θα πρέπει να μιλήσουμε για συνεταιρισμούς, συνεταιρισμούς για πωλήσει, αλλά και για ενεργειακές, ενεργειακοί συνεταιρισμοί, συνεταιρισμοί από τους πολίτες στην κοινωνία των πολιτών, καθώς και η δυνατότητά του, να, κατασκευ... να παράγουν ε, ανανεώσιμες ε, ενέργειες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν μέσα στα κτίρια. Αυτές είναι προτάσεις που θα υποβάλουμε εμεί ω πράσινοι μέσα στο πλαίσιο τη μεταρρύθμισης τη ενεργειακή και τη μεταρρύθμισης των ε, κτιρίων. Σας ευχαριστώ πολύ και τώρα από την ΚΟΕ ο κύριος Ηλικιώτης. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, ο στόχο που τίθεται για βελτίωση τη ενεργειακή απόδοση των κτηρίων είναι πολύ σημαντικό και μπορεί πραγματικά να αποφέρει πολλά ωφέλη για την κοινωνία εφόσον προωθηθεί σωστά με ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράση. Για την ομάδα μα στην QNGL αποτελεί προτεραιότητα να επιταχυθεί η ανακαίνιση για την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι που έχουμε θέσει για την προστασία του περιβάλλοντο και ταυτόχρονα επιτύχουμε τη βελτίωση τη υγεία των ανθρώπων που ζουν σε παλαιά χτίρια με βλαβερές κλιματικές συνθήκες. Με την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης όμως δεν θεωρούμε πώς μπορεί να καταπολεμηθεί η ενεργειακή φτώχεια όπως αναφέρεται η πρόταση της Κομισιόν. Για να πετύχουμε αυτό, την καταπολέμηση δηλαδή της ενεργειακής φτώχειας, χρειάζεται να ενισχυθεί η κοινωνική πολιτική, να προωθούν μέτρα που να διασφαλίζουν πραγματικά σε όλους ισότιμη και φτηνή πρόσβαση στην ενέργεια ως δημόσιο κοινωνικό αγαθό. Μπορεί όμω, σε κάποιο βαθμό η αύξηση τη ενεργειακή απόδοση στο κτηρίο να οδηγήσει στο να μειωθεί το κόστο για τα νοικοκυριά και αυτό θα είναι μια έστω και μικρή βοήθεια για τα 23 εκατομμύρια νοικοκυριό στην Ευρωπαϊκή Ένωση που ζουν σε συνθήκε ενεργειακή φτώχεια. Ιδιαίτερα προβληματική όμω κατά τη γνώμη μα είναι η λογική στην οποία προτείνεται από την Επιτροπή να στηριχτεί πρωτοβουλία για έξυπνη χρηματοδότηση για τα έξυπνα κτίρια επί της ουσίας θα χρησιμοποιεί εγγύησει του δημοσίου για να μοχλεύει ιδιωτικές επενδύσεις καθώς θα περιορίζει το ρίσκο των ιδιωτών. Κατ' επέκταση και πάλι δεν θα υπάρχει καμία εγγύηση πως οι επενδύσεις θα γίνονται εκεί που υπάρχει πραγματική ανάγκη αλλά και εκεί που θα επιλέγουν οι ιδιώτες επενδυτές. Εάν πραγματικά θέλουμε να λειτουργήσει προ όφελο τη κοινωνία η οδηγία για την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων, θα πρέπει να τεθεί ω προτεραιότητα η χρηματοδότηση των κτηρίων, των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, το κτηρίο σε υποβαθμισμένε και απομονωμένε περιοχέ, καθώ και το κτηρίο στι οποίε στηγάζονται μικρομεσαίε επιχειρήσει. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μάλιστα και τώρα ο κύριος Ταμπουράνο από το EFDD. Σε ευχαριστώ. Εμείς είμαστε πολύ, πολύ ε, ε, ευνοϊκά διακείμενοι σε αυτή την πρόταση, ιδιαίτερα όσον αφορά την ευθυγράμμιση με το θέμα της ε, ανανέωσης, ανακαίνησης των κτηρίων και την ε, ενεργειακή μεταρρύθμιση των κτίριων. Εκεί μπορούμε να δούμε περισσότερο τον αντίκτυπο της ε, ενεργειακής απόδοσης ε, γιατί ο ρυθμός ανανέωσης των κτιρίων είναι πολύ αργός και το να επικεντρωθούμε μόνο σε καινούργια κτίρια δεν θα δώσει μεγάλο αποτελέσμα. Είναι σημαντικό να δούμε την ανακαίνιση και ε, όσον αφορά τώρα την ε, ηλεκτρική κινητικότητα, είμαστε υπέρ. Θεωρούμε μάλιστα πως το 10% της προδιάθεσης ε, των πάρκων ηλεκτρικής κινητικότητας είναι ανεπαρκής. Και μάλιστα τα τελευταία νέα είναι ότι η Τέσλα θα λανσάρει στην αγορά ένα μικρό αυτοκινητάκι με κόστος 30.000 ευρώ. Οπότε ε, ε, αλλάζουν τα πράγματα στην ηλεκτρική κινητικότητα σε σχέση με το όσα ξέραμε μέχρι πριν από λίγους μήνες. Ε, τώρα, το smartness των κτηρίων επίσης να μετράται και να ενσωματωθεί και στα πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης όπως είμαστε υπέρ των συστημάτων ηλεκτρικής διαχείρισης που επιτρέπουν να ε, ωφέλει απτά για τους ε, ε, Κατοίκου των κτηρίων αυτών. Στο πακέτο αυτό το ενεργειακό θα πρέπει ποτέ να ξεχνάμε βέβαια τη γενικότερη εικόνα, το big picture. Γι' αυτό όσον αφορά τη διακυβέρνηση να πούμε ότι τα μακροπρόθεσμα σχέδια για την απόδοση της ενέργειας στα κτίρια θα πρέπει να ενταχθούν σε όλα τα προγράμματα τα εθνικά και θα πρέπει επίσης να ρυθμιστεί η παραγωγή των μεγαβάτ αυτών ώστε να μην υπάρχουν εξαιρέσεις, μονοπόλια ή κατάχρηση ε, κυρίαρχης θέσης της αγοράς. Ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Έχουμε και άλλους 12 ομιλητές, συναδέλφους μάλλον που θέλουν να συμβάλλουν σε αυτή τη συζήτηση. Ένα λεπτό έκαστος. Γκρίφιν πρώτα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Η απόδοση της ενέργειας είναι το πρώτο και καλύτερο καύσιμο. Ε, τώρα, όσον αφορά την ανανέωση των κτηρίων στην Ευρώπη, και τη... είναι τεράστιο το στόκ, αλλά τη... η πρόταση της Κομισιόν δεν ανταποκρίνεται στα εύρος του έργου. Εστιάζει περισσότερο στα FEE e κτίρια για την FEE e κατανάλωση και απόδοση. Το υποστηρίζω βέβαια αυτό, αλλά πιστεύω πως θα πρέπει να είμαστε το ίδιο ε, φιλόδοξοι μάλλον για την ανανέωση των ήδη υπαρχών των κτιρίων, ειδικά για τους ανθρώπους που ζουν στη φτώχεια και ζουν και στα λιγότερα αποδοτικά ενεργειακά κτίρια. Ε, γι' αυτό θα πρέπει να συμπεριληφθεί ένα συγκεκριμένο στόχο για τη βελτίωση τη απόδοση για τι εργατικέ κατοικίε και για ε, τις ε, κατοικίες με χαμηλή απόδοση. Αυτό θα σήμαινε βελτίωση της ευημερία των κοινοτήτων των κοινωνιών και θα τόνωνε και την οικονομία, ώστε να έχουμε 3 εκατομμύρια σπίτια που μπορούν να ανακαινιστούν και 7 εκατομμύρια κόσμος να βγει έτσι από την φτώχεια. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Βαν Μπρέμπτ. Ευχαριστώ πολύ. Ε, να κάνω κάποιες πολιτικές φύση ε, παρατηρήσει γιατί θα έχουμε την ευκαιρία να μπούμε στι λεπτομέρειε. Ε, όπως αναφέρθηκε από τον εισηγητή στην εισήγησή του, θα πρέπει να τονίσω ότι δεν είναι μόνο πολύ σημαντικό αυτό ο φάκελο, αλλά και δεν είναι μόνο το κομμάτι της Συνεργειακής Ένωση, αλλά είναι ε, υποχρέωσή μα για να ανταποκριθούμε στη Συμφωνία του Παρισιού. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και το υπογραμμίζω γιατί δεν μπορεί κανεί να διαλέξει κάτι από όλα αυτά. Θα πρέπει να το δούμε ω μια γενική δέσμευση. ETS, καθαρή ενέργεια, μεταφορέ, όλα μαζί. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε λοιπόν και να έχουμε αυτήν την γενική εικόνα και να μην αφήσουμε αυτά τα ζητήματα εκτός. Δεύτερον, παρατήρηση που έγινε και από άλλους ότι θα πρέπει να ε, έχουμε και να τονίσουμε τα ωφέλη από αυτούς τους στόχους. Ε, η ενέργεια και η απόδοση μπορεί να δημιουργήσει πάρα πολλές θέσεις απασχόλησης. Θα μπορέσουμε έτσι να καλύψουμε τη φτώχεια στην ενέργεια. Πολύ συγκεκριμένε δεσμεύσεις λοιπόν ε, αναλαμβάνουμε μέσω αυτής της πρότασης. Ευχαριστώ ο κύριος Κέλλη. Σας ευχαριστώ πολύ. Πρέπει να πω καταρχάς κύριος, ε, ότι ο κύριος Μπένσεν είναι εισηγητής, αυτό με χαροποιεί ιδιαίτερα γιατί είναι ειδικό στο θέμα, αλλά είναι και ο ίδιος υπόδειγμα γιατί έχει ανακαινήσει το ίδιο του το σπίτι με τέτοια στάνταρα ε, ενεργειακής απόδοσης. Κάτι που δεν αναφέρθηκε μέχρι στιγμής είναι το θέμα της παιδείας. Επειδή εγώ προέρχομαι από την Ιρλανδία, ε, και ζήσαμε και τη φούσκα την οικοδομική όπου χτίστηκαν ε, χιλιάδες σπίτια όπως όπως. Δεν θέλω να συμβεί ξανά αυτό το πράγμα σε καμιά χώρα. Εφόσον μιλάμε για αποδοτικά ενεργειακά σπίτια θα πρέπει να είμαστε βέβαιοι πως ε, οι χτίστες, ε, οι εργολάβοι, οι υδραυλικοί, οι ηλεκτρολόγοι και όλοι να είναι ειδικοί για να το κάνουν σωστά αυτό. Το να λέει κανείς ότι είναι ειδικό δεν αρκεί. Σίγουρα λοιπόν εδώ θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι όσοι κάνουν αυτού του είδους τις ανακαινήσεις να είναι και ειδικά καταρτισμένοι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Επόμενος ομιλητής. Ε, πρόεδρε, γνωρίζουμε ότι τα κράτη-μέλη εν γέννη είναι υπέρ αυτής της ε, ε, ανανέωσης, αλλά πρέπει να μιλήσουμε όχι μόνο για τα σημαντικά θέματα, αλλά και για τις λεπτομέρειες. Αν υπάρξει σύγκρουση με το Συμβούλιο, θα τραβήξει πολύ η ιστορία και αυτό θα καθυστερήσει την εφαρμογή. Όσον αφορά την οδηγία, είναι αλήθεια ότι δεν αλλάζει πραγματικά την... Ε, ε, την διατύπωση, αλλά εξακολουθώ να πιστεύω πως υπάρχουν κάποια ζητήματα. Καταρχάς, ο ορισμός της, των κτηρίων μηδενικής κατανάλωσης λείπει. Αφήνεται αυτό στην καλή θέληση των κρατών μελών, πράγμα που πιστεύω δεν είναι καλή ιδέα. Οι απαιτήσει για αυτού το είδους τα κτηρία θα πρέπει να ορίζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η αναθεωρημένη οδηγία περιλαμβάνει το αρχικό άρθρο 4 ε, της οδηγίας περί ενεργειακής απόδοσης, το οποίο καλωσορίζω γιατί αυτό μπορεί να βοηθήσει επίση στη χρηματοδότηση τη ανακαίνιση της κτηρίων και στη μείωση του στόχη. Καλό θα ήταν όμω να βγει και η, το άρθρο 5 εδώ και από την πραλιά οδηγία για να μην καλύπτονται μόνο τα κυβερνητικά κτίρια αλλά όλα τα δημόσια κτίρια. Μάλιστα, ο κύριο Κόχλιτσεκ. Ευχαριστώ. Ε, νομίζω πως τα δημόσια κτίρια και οι εργατικές κατοικίες θα πρέπει να αποτελέσουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση και την μόνωση. Δεν μιλάμε όμως μόνο για μόνωση, αλλά και για σκίαση, διότι ειδικά στα νότια μέρη του, της Ευρώπης θα πρέπει να μπορούμε να εξοικονομήσουμε περισσότερη ενέργεια εάν προβλέψουμε σωστή σκίαση των κτηρίων αλλά και εξαιρισμό. Εάν ένα κτίριο είναι καλά ε, μονομένο πρέπει να εξαιρίζεται και σωστά γιατί διαφορετικά δημιουργείται ένα μικροκλίμα το οποίο είναι πολύ ζωφερό για τον κόσμο που κατοικεί σε αυτά τα αεροστεγή κτίρια. Απλή τρόποι λοιπόν αξιολόγησης ε, των ε, τεχνικών, εάν θέλουμε λοιπόν να μονώσουμε τα υπάρχοντα κτίρια χρησιμοποιώντας ευρωπαϊκά χρήματα και μειώνοντας την ενεργειακή φτώχεια, η απάντηση είναι η, το καθολικό δικαίωμα για μήνυμο πρόσβαση στην ενέργεια. Τελευταίο μου σχόλιο είναι ότι αν θέλουμε να έχουμε ηλεκτρική, ηλεκτρονική κινητικότητα θα πρέπει να εναρμονίσουμε και τις βρίζες. Γιατί αυτή τη στιγμή είναι σχεδόν αδύνατον να, ε, να φορτίσει κανείς το τηλέφωνο του παντού. Ο κύριος Ευχαριστώ πολύ, Μπεν. Σε ευχαριστώ πάλι πάρα πολύ για την πρώτη σου αυτή θετική δήλωση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε ένα σημαντικό σχεδιασμό και όντω υπάρχει απόκληση αυτή τη στιγμή ανάμεσα στην ευρωπαϊκή και τι εθνικέ νομοθεσίε. Α ξαναδούμε λοιπόν το κείμενο αυτό που έχουμε επιτάπητο, για να δούμε τελικά αν η πτυχή των κοινωνικών εργατικών κατοικιών μπορεί να αποτελέσει τμήμα τη μακροπρόθεσμη στρατηγική αν δούμε τι γίνεται σε πάρα πολλές χώρες, τι έγινε αυτό το χειμώνα, όπου υπήρχαν πάρα πολλές χώρες που φτάσανε σε πάρα πολλά υψηλά επίπεδα ατμοσφαιρικής ρήπανσης. Υπήρχαν πάρα πολλέ χώρε που αντιμετώπισαν πολλά τέτοια προβλήματα. Νομίζω θα πρέπει να έχουμε μια σχετική στρατηγική και για αυτό το ζήτημα. Μπέντ, υπάρχει ένα άλλο ζήτημα, επί το οποίο δεν ξέρω αν έχει βρεθεί κάποια λύση. Οι τιμέ του πετρελαίου και οι τιμέ του φυσικού αερίου είναι πλέον αρκετά χαμηλέ και οι προβλέψεις του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας και άλλων σχετικών οργανισμών θα παραμείνουν χαμηλές οι τιμές αυτές. Πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε λοιπόν ένα επιχειρηματικό μοντέλο βάσει του οποίου θα χρησιμοποιηθούν ιδιωτικά κεφάλαια σχετικά με τις τιμές αυτές φυσικού αερίου και πετρελαίου προκειμένου να καταφέρουμε τελικά στα πλαίσια του ε, κτηριακού το που έχουμε να φτάσουμε σε μηδενικές εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα και να καταφέρουμε κατά αυτόν τον τρόπο να δημιουργήσουμε συνθήκες θετικής μόχλευσης όσον αφορά τα ιδιωτικά κεφάλαια. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να ασχοληθούμε λίγο περισσότερο με αυτό. Πώ μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε καλύτερα αφενό μεν του δημόσιου πόρου, αλλά καθώ αυτή τη στιγμή οι τιμέ διοξιδίου του άνθρακα, οι τιμέ πετρελαίου και φυσικού αερίου είναι χαμηλέ, δεν νομίζω ότι μπορούμε να προσελκύσουμε πάρα πολλέ επενδύσει μόνο από τα ιδιωτικά κεφάλαια όσον αφορά την ανακαίνιση των κτηρίων. Νομίζω ότι και το ζήτημα αυτό πρέπει να σα απασχολήσει. Πρόεδρο, ευχαριστούμε. Ο κύριο Μπλάνκο Λόπε έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Η ενεργειακή απόδοση των κτηρίων είναι ουσιώδηση στη στρατηγική ε, μείωση της χρήσης του άνθρακα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, ε, πρέπει λοιπόν και να προσέξουμε ε, ε, γιατί υπάρχει μεγάλο περιθώριο ε, κέρδους. Έχουμε λοιπόν πρόβλημα με τα κτίρια κατά 70%. Δεν είναι ενεργειακά αποδοτικά τα κτίρια. Γνωρίζουμε ότι ε, οι καινούριε ενέργειε είναι πιο αποτελεσματικές και πιο φθηνέ. Μάλιστα, αυτό θα σημάνει κατανάλωση λοιπόν λιγότερης ενέργειε, με προώθηση της άνεσης και θα προωθήσει και τις θέσεις απασχόλησης. Ε, πολλές ευκαιρίες για τα καταπολέμηση της ενεργειακή στόχιας, δε, από την οποία υποφέρουν 23 εκατομμύρια οικογένειες στην Ευρώπη. Είναι σημαντικό να, τον, να, να προωθηθούν αυτές οι πληροφορίες, βελτιώνοντας τα πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης, βελτιώνοντας τον εντοπισμό μέτρων με τρόπο αποδοτικό και μέσω των απαραίτητων υποδείσεων. Είναι μια ευκαιρία λοιπόν που έχουμε μπροστά μας. Ευχαριστούμε πολύ. Η κυρία Σπυράκη έχει το λόγο. Σα ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Είμαι και εγώ ευτυχή που είναι ραπορτέρο ο κύριο Μπένσον, διότι το δικό του έξυπνο σπίτι είναι ενδεχομένω ένα υπόδειγμα. Αλλά θα ήθελα να πω ότι εδώ είμαστε για να γεφυρώσουμε την απόσταση ανάμεσα στο έξυπνο σπίτι του κύριου Μπένσον και στα παλιά φτωχά σπίτια και κτίρια, στα οποία ζουν χιλιάδε άνθρωποι στην Ευρώπη. Σύμφωνα με βρήματα έρευνα που διενεργήθηκε με πρωτοβουλία μου στο πολυδομικό συγκρότημα τη Θεσσαλονίκη, 6 στα 10 νοικοκυριά δυσκολεύονται να πληρώσουν το ηλεκτρικό ρεύμα ενώ 14% των οικογενειών αυτών ζει μια περίοδο χωρίς καθόλου ηλεκτρικό ρεύμα. Το 13% του εισοδήματο είναι η μέση δαπάνη για την ενέργεια στο πολυδομικό σκρότημα τη Θεσσαλονίκη, όταν ο καταρχήν ορισμό για την ενεργειακή φτώχεια δείχνει ότι ενεργειακά φτωχό είσαι αν ξοδεύει πάνω από το 10% του εισοδήματό σου. Τι προτείνω. Καταρχήν ενθάρρυνση των κρατών μελών για τη δημιουργία χρηματοδοτική πλατφόρμα που σε συνδυασμό με τους πόρους του ΕΨΥ, του σχεδίου Juncker, των διαρθρωτικών ταμείων, αλλά και των ταμείων που έρχονται από τον ιδιωτικό τομέα, θα μπορέσουν να αναλάβουν αυτό το γιγάντιο έργο. Δεύτερο, ενημέρωση. Ενημέρωση των φτωχών ανθρώπων για τα απτά ωφέλη που θα έχουν. Είτε με τη μείωση του λογαριασμού, είτε με τη βελτίωση της καθημερινότητάς τους, είτε και με τα δύο. Σας ευχαριστώ. Thank you very much. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Δεν θα ήθελα να επαναλάβω αυτά που είπαν οι συνάδελφοι, τα οποία τα βρήκα πολύ πιστικά. Νομίζω πάντως ότι ένα από τα στοιχεία, τα λιγότερα θετικά υποσχόμενα της πρότασης αυτής, είναι το να έχουμε μία απλή αναδιατύπωση εδώ πέρα. Δεν έχουμε πραγματική αναθεώρηση εδώ πέρα τις οδηγίες όπως θα έπρεπε να έχουμε. Αυτή τη στιγμή, μέσω της πρότασης αυτής, πραγματικά δεν καταφέρνουμε να κάνουμε ενεργειακή εξοικονόμηση, όπως λέγεται στο άρθρο 7 της ε, οδηγίας 31-2010 ε, για την ενεργειακή απόδοση. Γίνεται εδώ μια παράταση απλώς νεφιστάμενων διατάξεων. Υπό το φως ε, των όσων έχει πει το Κοινοβούλιο, μήπως θα έπρεπε να ήμασταν πιο φιλόδοξοι δηλαδή να αναθεωρηθούν προς τα πάνω οι αρχικοί στόχοι, γιατί μέσω της ε, εξοικονόμησης προβλέπεται 1,25% προς τους τελικούς χρήστες, ουσιαστικά επαναλαμβάνουμε τα όσα είχαμε κάνει στο παρελθόν. Επίσης, θα πρέπει να επεκτεθεί το πεδίο εφαρμογή έτσι ώστε να καλύπτονται και άλλα κτίρια, όπως και τα δημόσια κτίρια, για παράδειγμα. Κατά αυτόν τον τρόπο μπορούμε να έχουμε μια μεγαλύτερη, αν θέλετε, διοικητική συνέπεια στα όσα νομοθετούμε. Και επίσης μπορούμε κατά αυτόν τον τρόπο να πετύχουμε μια ενεργειακή απόδοση όλων των κτηρίων που θα πρέπει να είναι βασικός στρατηγικός μας στόχος. Ευχαριστούμε πολύ. Κάριντς. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όντω είναι πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση αυτή. Να τονίσω κάτι από πρακτικής πλευράς. Είναι προφανές ότι ε, Μπορούμε όντω να αυξήσουμε την ενεργειακή απόδοση στα κτίρια, μπορούμε να εφαρμόσουμε φιλοπεραβαλλοντικέ πολιτικές. Υπάρχει το ζήτημα πάντως του κόστους και το ζήτημα της ε, αποκατάστασης των κτηρίων. Βλέπετε εδώ πέρα ότι έχουμε το παράδειγμα των τριών βαλτικών χωρών, αλλά έχουμε και πολλές χώρες από την κεντρική και ανατολική Ευρώπη, οι οποίες έχουν πολλά σοβιετικά κτίρια από τη δεκαετία του 70 και του 80, οι οποίες, τα οποία κτίρια δεν είναι ενεργειακά αποδοτικά. Κανείς δεν ενδιαφερόταν από την εποχή εκείνη για την ενεργειακή απόδοση. Προκειμένου λοιπόν να ανακαινήσουμε τα κτίρια αυτά, θα πρέπει πραγματικά να δούμε αν υπάρχουν οι απαραίτητες δεξιότητες για να γίνει αυτή η ανακαίνιση. Η μόνωση ενός κτίριου δεν σημαίνει ότι θα βάλουμε απλώς μονοτικό υλικό. Γιατί αν κάνετε μόνο αυτό το πράγμα, τότε δεν θα υπάρχει καλή κυκλοφορία του αέρα. Αν δεν προβλέψετε και ένα σύστημα αερισμού του κτιρίου Αν απλώς ενισχύσετε τη μόνωση, τότε ενδεχομένω το κτίριο αυτό να μην λειτουργεί κανονικά και να είναι ανθυγιεινό. Καταλαβαίνετε όμως ότι ε, όλα αυτά επιφέρουν ένα κόστος. Τα περισσότερα κτίρια στις χώρες μας αυτά δεν είναι κοινωνικά ή εργατικά κτίρια. Καταλαβαίνετε ότι ε, στα κτίρια αυτά κατοικούν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι έχουν ε, χαμηλά εισοδήματα, οι περισσότεροι άνθρωποι που έχουν υψηλότερα εισοδήματα ουσιαστικά βρίσκονται ήδη σε κτίρια τα οποία είναι πολύ πιο ενεργετικά αποδοτικά. Οι άνθρωποι λοιπόν αυτοί όντας φτωχοί μένουν σε κτίρια τα οποία δεν είναι εργατικές κατοικίες και καλούνται να επιβαρυνθούν αυτοί με το κόστος ανακαίνιση των κτιρίων τους. Αυτό προφανώς πρέπει να αποφευχθεί. Ευχαριστούμε πολύ, λέει Πρόεδρος. Θα ήθελα να αφαιρθώ σε αυτά που είπε ο κύριο Κέλλη, ο οποίο είπε ότι ο κύριο Μπένσεν έχει ένα καταπληκτικό σπίτι, το οποίο είναι παράδειγμα προ μίμηση. Να σα υπενθυμίσω ότι ε, οι σκιώδεις ηγητέ, και απευθύνομαι στους σκιώδεις ηγητέ, ότι ο μεγαλύτερος ιδιοκτήτης κτηρίων στα 28 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι οι κυβερνήσεις. Πρέπει λοιπόν και οι κυβερνήσεις με τα δικά τους κυβερνητικά δημόσια κτίρια να δώσουν το θετικό παράδειγμα. Αναφέρθηκε ο κύριος Χάριν σε κτίρια τα οποία βρίσκονται σε αισχρή κατάσταση. Πολύ συχνά τα κτίρια αυτά Δυστυχώς είναι δημόσια κτίρια. Κάθε φορά λοιπόν που θέλουμε να επιβάλλουμε εμεί κανονισμού στον ιδιωτικό τομέα, α μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και ο δημόσιο τομέα, ο οποίο καλείται αυτή τη στιγμή να αναλάβει τι ευθύνε του. Θα λέει λοιπόν στον εισηγητή ότι θα πρέπει κάπου να συμπεριλάβει στην έκθεσή του ότι ο μεγαλύτερο ιδιοκτήτη κτηρίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το ίδιο το δημόσιο. Ο κύριο Γκέρεκ έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αναφερθήκαμε στην ενεργειακή απόδοση των κτηρίων εκτενέστατα. Θα πρέπει όμως να έχουμε κατά νου ότι το ζήτημα αυτό πολλές φορές είναι απλώς τοπικό ζήτημα, διότι η θέρμανση, όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορεί να ταξιδέψει μεγάλες αποστάσεις και υπάρχουν και μεγάλες αποκλήσεις και διαφορές στην Ευρώπη όσον αφορά τις ε, γεωγραφικές συνθήκες που ισχύουν. Στις βόρειες χώρες ε, χρειαζόμαστε 200, 200 κιλοβατόρες ενώ 30 κιλοβατόρε μπορεί για παράδειγμα να αρκούν σε κάποιες χώρες της Νότιας Ευρώπης. Δεν νομίζω λοιπόν ότι μπορούμε να έχουμε εδώ πέρα ένα ομοιόμορφο σύστημα το οποίο θα μπορούσε να ισχύσει για όλες τις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά για παράδειγμα τις ανάγκες θέρμασης των κτηρίων. Πρώτον αυτό, δεύτερον. Το εγχείρημα είναι τεράστιο αυτή τη στιγμή για τους πολιτικούς μηχανικούς, για τους αρχιτέκτονες στα διάφορα κράτη-μέλη το εγχείρημα αυτό θα πρέπει αυτοί να το αναλάβουν και νομίζω ότι θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν καλύτερα και οι ίδιες οι κλιματικές συνθήκες που υφίστανται στα διάφορα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζω ότι κατά αυτόν τον τρόπο μπορούμε όντως να έχουμε την καλύτερη δυνατή ενεργειακή απόδοση των κτηρίων. Ο κύριος Ρόλ έχει το λόγο. Όλοι είπαμε πόσο σημαντική είναι η εξοικονόμηση ενέργειας και πόσο κακή είναι η ενεργειακή φτώχεια. Αλήθεια είναι όλα αυτά. Τι μπορούμε όμως να κάνουμε. Να πω ένα πράγμα. Αν ε, αναβαθμίζουμε τις διατάξεις για τα κτίρια, αυτοί που κατασκευάζουν κτίρια θα χρησιμοποιούν περισσότερα χρήματα. Θα είναι πιο ακριβά τα κτίρια. Δεν θα μπαίνουν μέσα ε, ε, εκεί λοιπόν άνθρωποι που δεν μπορεί να πληρώσουν τα ακριβά νίκια. Και αυτό σημαίνει ότι θα είναι αντικίνητρο για κατασκευή τέτοιων κτιρίων αφού το κόστος θα είναι τόσο μεγάλο και επειδή έχουμε τόσο πολύ ε, απαιτητικές ε, αλλά και ε, δαπανηρές διατάξεις. Αυξάνομαι το κόστος, δεν κατασκευάζονται λοιπόν κτίρια ή δεν μπορούν να κατοικηθούν και να χρησιμοποιηθούν από το μέσον όρο. Ε, φτάνουμε λοιπόν παρόλες τις καλές προθέσεις στο αντίθετο αποτέλεσμα από αυτό που επιδιώκουμε. Ευχαριστώ. Ο κύριος Νίκα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε ένα σχόλιο. Πρέπει να έχουμε κάποια υποχρεωτικά στοιχεία στην ευρωπαϊκή πολιτική. Στις ανατολικές χώρες υπάρχουν μεγάλα ε, συγκροτήματα ε, διαμερισμάτων και για να ανακαιτινιστούν για την ενεργειακή απόδοση θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν περιφερειακά κονδύλια. Υπάρχει, ε, το προβλέπει η Γενική Διεύθυνση Ρέτζιο, αλλά δεν καλύπτονται από εκεί οι πρωτοβουλίε των τοπικών κοινοτικών δημοτικών συμβουλίων. Να καλύπτονται δηλαδή από κονδύλια κοινοτικών ε, ε, συμβουλίων. Επίσης, είναι πολύ δύσκολη η διαδικασία λήψη των αποφάσεων, γιατί ε, σε μια συνέλευση και ένα να διαφωνεί δεν μπορεί να προχωρήσουν οι αποφάσει. Καμιά φορά δηλαδή υπάρχουν καλέ πρωτοβουλίε που μπλοκάρονται από τη γραφειοκρατία. Και αυτά όλα ε, δεν ε, προβάλλονται και δεν επιλύονται. Άρα δεν χρησιμοποιούνται ενωσιακά κονδύλια και δεν έχουμε και κτίρια με σωστή ενεργειακή απόδοση. Ευχαριστώ πολύ. Ε, κύριε Νίκα. Άλλος που να θέλει να λάβει το λόγο, δεν βλέπω κανέναν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ε, εξαιρετική πειθαρχία. Ο κύριος Χότσεν από τη Γενική Διεύθυνση Ενέργειας θα μας ε, μιλήσει τώρα. Ευχαριστώ. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση ήδη από τώρα και προσβλέπουμε στη συνέχειά της. Ε, στον κύριο Μπέντσεν θα ήθελα να πω ότι περιμένουμε να ακούσουμε περισσότερα για τις ιδέες σας και πώς η νομοθεσία μπορεί να προωθήσει την πρόσβαση στην ε, ιδιωτική χρηματοδότηση. Ε, θα πρέπει να γίνουν κάποια πράγματα νομοθετικά. Ακούσαμε με ενδιαφέρον αυτά που είπατε. Και επίσης ε, πώς θα αποφύγουμε τα προβλήματα της ηλεκτρονικής κινητικότητας. Στην κυρία Κουμπούλα Νάντρο και στον κύριο Κέλλη θα πω ότι ναι, συμφωνούμε ότι χρειάζεται να επικεντρωθούμε στα προσόντα από το Horizon 2020 ε, που έχει ένα πρόγραμμα, μια συνιστόσα για ε, απόκτηση περισσότερων προσόντων. Δουλεύουμε πάνω σε αυτό στην πράξη. Ε, χρειάζεται δηλαδή εδώ παράλληλη δράση με την νομοθεσία. Στον κύριο Τσάτσακο που μίλησε για το κόστος της ηλεκτρονικής κινητικότητας. Υπάρχει ένα κόστος, το έχουμε εκτιμήσει. Έχουμε, είναι περίπου 80 δις για τα κτίρια που δεν είναι κατοικίες. Παραλληλά ε, έχουμε το πρόβλημα της κότας και του αυγού στην ηλεκτρονική κινητικότητα. Αν δεν κάνουμε αυτή την παρέμβαση δεν μπορούμε να ε, ασκήσουμε επιρροή διαφορετικά. Θα πρέπει να δούμε πού γίνεται η χρέωση θα πρέπει λοιπόν να βεβαιωθούμε ότι θα είναι αποδοτική η επένδυση. Ε, να έχουμε δηλαδή το καλύτερο, την καλύτερη σχέση κόστους ωφέλειας. Για τις μονοθυριδικές υπηρεσίες συμφωνούμε και στα πλαίσια του Horizon 2020 θα κοιτάμε αυτά να, ε, και σε εθνικό επίπεδο δηλαδή να δούμε πώς θα λειτουργήσουν όλα αυτά για τη χρηματοδότηση έξυπνων κτηρίων στη χώρα σας κάποιες ιδιωτικές εταιρείες έχουν κάνει πολύ αποτελεσματικά προγράμματα. Καλό είναι να βρουν μιμητές και σε άλλα κράτη-μέλη. Θα το δούμε αυτό πιο καλά. Συμφωνούμε με τον κύριο Ματσελέζη σχετικά με την σύνδεση με το ευρύτερο σύστημα. Ένας ρόλος του δίκτυου ευφυΐας ε, ε, ε, είναι ότι δείχνει αν μπορεί να υπάρξει σύνδεση σε ένα ευρύτερο δίκτυο και αν μπορούν ε, να ε, αξιοποιηθούν οι χαμηλότερες τιμές ενέργειας σε ένα κτίριο ενεργειακής απόδοσης, εκμεταλλευόμενο ηλιακή ενέργεια κλπ. όταν υπάρχει ηλιοφάνεια. Αυτό είναι σημαντικό να το λάβουμε υπόψη μας. Δεν μας νοιάζει μόνο ε, να βρούμε λύσεις υψηλής τεχνολογίας, ένα κτίριο το οποίο έχει μια δεξαμενή για θερμό νερό ε, που μπορεί να ε, θερμανθεί όταν υπάρχει ηλιοφάνεια. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό και είναι και μια απλή λύση. Δεν είναι μόνο οι λύσεις υψηλής τεχνολογίας που μας πάνε μπροστά. Στον κύριο Σιλικιώτη να πω για την ενεργειακή φτώχεια, δηλαδή αυτό το είπαν και πολλοί άλλοι παρεμβαίνοντες. Ε, εμείς λέμε ότι ήδη από αυτά τα προγράμματα ωφελούνται τα χαμηλά εισοδήματα όταν νοικιάζει κανείς ένα κίνητο θα πρέπει να ενημερωθεί ε, ο ενοικιαστής ε, για την ενεργειακή απόδοση. Θα κάνει τους λογαριασμούς του και θα δει τι θα πληρώνει. Αν είναι ανακαινισμένο το κτίριο πρέπει να βελτιώσει την ενεργειακή απόδοση. Αυτοί που νοικιάζουν σπίτια και αυτοί που είναι ιδιοκτήτες όλοι θα ωφεληθούν από αυτές τις επενδύσεις. Γι' αυτό Κάνοντας αυτό και μόνο βλέπουμε ότι 3 εκατομμύρια νοικοκυριά βγαίνουν από την φτώχεια. Ε, ε, αυτό δεν σημαίνει, γιατί ε, βρίσκονται απλές λύσεις σε, ένα πρώτο επίπεδο. μόνο και μόνο που κινούμεθα προς αυτή την κατεύθυνση ωφελούμε και τους φτωχούς. Κύριε Ταμπεράνο, και κύριε Τούρμες υπάρχουν συνδέσεις με τον σχεδιασμό της αγοράς, τη διακυβέρνηση και την ανανεώσιμη ενέργεια γιατί πολλά από αυτά που κάνουμε εδώ αξιοποιούν την οδηγία ε, ενεργειακής απόδοσης όχι μόνο για, να, για, την ενεργειακή απόδοση ως αυτό σκοπό αλλά και για να προωθήσουμε τις ανανεώσιμες πηγές. Ε, τα μακροπρόθεσμα σχέδια ε, έχουν σχέση και σύνδεση με τη διακυβέρνηση. Δηλαδή, όταν τα Υπουργεία κάνουν τον ε, μακροπρόθεσμο ενεργειακό του σχεδιασμό, πρέπει να ξέρουν ε, τι συμβολή μπορεί να έχουν στον σχεδιασμό αυτό τα κτίρια και η ενεργειακή τους απόδοση. Η σύνδεση με το Παρίσι και εδώ και αυτά και άλλα μέτρα θα αποτελέσουν κομμάτι της συμβολής της Ένωσης στο να δούμε πώς θα συμβάλλουμε στις υποχρεώσεις που αναλάβαμε και μετά τις το, 2030. Ε, ένας τομέας που εδώ ε, έχουμε επιφυλάξει είναι το να διευρύνουμε το πεδίο εφαρμογής της πρότασης προσοχή μεγάλη εδώ. Δεν προτείναμε να δούμε τα ε, κτίρια σχεδόν μηδενικής ενεργειακής απόδοσης και δεν προτείναμε να μεταφέρουμε το άρθρο 5 ε, σε αυτή την πρόταση, εκείνο από τα, κεντρικά, τα ε, κτίρια της κεντρικής κυβέρνησης, γιατί δεν έχει νόημα να κάνουμε διεύρυνση για να συμπεριλάβουμε τον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Και ο κίνδυνος ε, του να ανοίξουμε κι άλλες διατάξεις είναι, και νομίζω ότι συζητήσαμε για το ότι πρέπει να τα βρούμε και με το Συμβούλιο. Δεν θέλουμε να περιπλέξουμε τις συζητήσεις και να τις επιμικίνουμε σε τομείς όπου δεν χρειάζεται. Το πεδίο εφαρμογής θα πρέπει να μείνει εκεί που το έχουμε βάλει εμείς. Τώρα για τα δημόσια κονδύλια το θέμα του κυρίου Τούρμες. Βέβαια μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει ε, κρατικά κονδύλια, δημόσια κονδύλια. Κι άλλα όμως μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Αυτό μπορεί να γίνει αν βελτιώσουμε το πλαίσιο και βελτιώσουμε ε, την κατάσταση ώστε να μειωθούν τα εμπόδια. Επίσης στα έξυπνα κτίρια χρησιμοποιείται μια σειρά δεδομένων σχετικά με τον αντίκτυπο των ε, παρεμβάσεων, αν αλλάξει ένα παράθυρο τι πόσο υπολογίζουμε ότι μειώνεται η, η, αναβαθμίζεται η απόδοση ούτως ώστε να υπάρχει μια βάση δεδομένων σχετικά με τις εξοικονομήσεις που μπορούν να γίνουν και αυτό να χρησιμεύσει και στο μέλλον. Ο κύριος Κάριν, ο κύριος Νίκα μίλησε για ε, συγκροτήματα κατοικιών ε, με ιδιώτες ιδιοκτήτες. Πολλές φορές ε, ε, είναι δύσκολο να βρεθεί συμφωνία για να γίνει μια ανακαίνιση και λοιπά στις γενικές συνελεύσεις δηλαδή των πολυκατοικιών καμιά φορά αν ένας διαφωνεί όπως είπατε δεν γίνεται τίποτε υπάρχουν όμως ε, τρόποι για να λυθεί το πρόβλημα και να γίνουν οι ανακαινήσεις ε, μπορούμε εδώ να χρησιμοποιήσουμε το παράδειγμα των δημοσίων κτηρίων και πως αυτά ε, αντιμετωπίστηκαν στη Λιθουανία να λύσουμε διδάγματα από εκεί. Τέλος, κύριε Ρόιλ, συμφωνούμε ότι πρέπει να κοιτάξουμε το κόστος. Όταν μιλάτε για νέα κτίρια, εδώ βλέπουμε πολύ πρόοδο στη, από τη σύγκληση ε, των, του κόστους ε, κτιρίων υψηλής ενεργειακής απόδοσης και λιγότερο υψηλής. Κάποια στιγμή θα πρέπει να γίνει μια ε, οικονομική επιλογή και μπορεί να ε, ε, έχουμε κίνητρα για να κάνουμε επιλογή κτηρίων σχεδόν μηδενικής ε, ενεργειακής κατανάλωσης. Αυτά προς το παρόν. Ευχαριστώ πολύ. Εντυπωσιακό. Καλύψατε σχεδόν κάθε ερώτηση. Τώρα ξαναγυρίζουμε στον εισηγητή, τον κύριο Μπένσεν, για να κλείσει το θέμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για όλα τα σχόλια από τους σκιώδες, τους συναδέλφους που ενδιαφέρονται για το φάκελο αυτό. Τα νέα κτίρια είναι 1,5% των, όλων των κτιρίων ετησίως. Πρέπει λοιπόν να εστιάσουμε στην υφιστάμενη μάζα κτιρίων. Ο μακροπρόθεσμος σχεδιασμός στα κράτη-μέλη είναι πολύ σημαντικός ε, εδώ και πολλοί συνάδελφοι σήμερα ανέφεραν την ενεργειακή φτώχεια και την ανάγκη ανακαινήσεων των δημοσίων κτιρίων και των ε, κατοικιών. Συμφωνώ με τον πρόεδρο ε, που σήμερα αναφέρθηκε σε πολλούς δήμους, κοινότητες, περιφέρειες, κράτη και είπε ότι έχουν πολλά ανεπαρκή ε, κτίρια. Να τονίσω σε αυτή τη φάση ότι είναι καλό ότι έχουμε το ΕΦΣΙ, έχουμε την ΕΤΕΠ, έχουμε διαρθρωτικά ταμεία κλπ αλλά τα δημόσια κονδύλια δεν λύνουν τις απαιτήσεις μας. Πρέπει να ε, βρούμε και ιδιωτική χρηματοδότηση. Αυτό είναι ένα κέριο ζήτημα που θα κρίνει την επιτυχία του φακέλου αυτού. Όλα πρέπει να τα εξετάσουμε και να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να προσελκύσουμε ιδιωτικές επενδύσεις. Επίσης, δεν είμαστε μόνοι μας. Ε, η ανανεώσιμη ενέργεια, τα θέματα διακυβέρνησης είναι πολύ σημαντικά και έχουμε σύνδεση με αυτά. Τέλος, πολύ σημαντικό, να ευχαριστήσω τον κύριο Χάρτσε και το, τους ε, συνεργάτες του για την εξαιρετική συνεργασία και περιμένω με μεγάλο ενδιαφέρον τις επόμενες διαπραγματεύσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ και τώρα θα περάσουμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης που είναι το υπαριθμό 11, προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι έχουμε μία ώρα προβλέψει για την έκθεση αυτή για τον εισηγητή του Σκιώδης και τη συζήτηση και θα δώσω τώρα το λόγο στον εισηγητή, τον κύριο Μπλάνκο Λόπεθ, για πέντε λεπτά. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Η πρόταση που υπέβαλε η Κομισιόν προσφέρει την ευκαιρία να προσεγγίσουμε την απαραίτητη προσαρμογή στις ε, αλλαγές της παραγωγής ε, ε, στον κόσμο της ενέργειας από την προηγούμενη νομοθεσία. Αυτό το νομοθετικό πλαίσιο θα πρέπει να περιλαμβάνει και να καλύπτει και τις, την πρόοδο της τεχνολογίας. Καταρχάς, θα πρέπει να σέβεται το δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών, πράγμα που είναι πολύ βασικό. δεύτερον, η σημαντική ανάπτυξη της αγοράς των ανανεώσιμων πηγών είναι σημαντική ευκαιρία για τις επιχειρήσεις μας αλλά και για την ε, δημιουργία θέσεων απασχόλησης, πράγμα που δεν μπορούμε να αφήσουμε κατά μέρος. Ε, θα πρέπει να αναπτύξουμε ε, ρόλο κλειδί στην ανάπτυξη των τεχνολογιών, να μιλήσουμε για μια βάση τεχνολογικής ανάπτυξης και να συζητήσουμε με ειδικούς ε, του χώρου. Επίσης, η τιμή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ε, είναι τόσο χαμηλή και επιτρέπει ότι να μην χρειάζεται να ανησυχούμε για την οικονομική βιωσιμότητα αυτής της εξέλιξης. Αντίθετα, πρόκειται για ευκαιρία για να έχουμε αυθινή ενέργεια που θα μας επιτρέψει να έχουμε και ανεξαρτησία ενεργειακή και να έχουμε πιο ανταγωνιστική βιομηχανία. Να έχουμε λοιπόν ε, τέτοια στοιχεία μέσα σε αυτή την πρόταση. Αυτό είναι όντως ε, αλήθεια, όμως έχουμε την ε, αίσθηση ότι δεν είναι αρκετέ αυτέ οι προτάσει σε σχέση με το μέγεθο των στόχων. Πιστεύω ο στόχο ε, του Κοινοβουλίου θα πρέπει να είναι να επιφέρει συνοχή στους στόχους που έχουμε ορίσει για το 2030 και αυτούς που έχουμε στέσει για το 2050. Γι' αυτό ο στόχος ε, για τη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο 27% ε, θα επιτρέψει και την μείωση της χρήσης του, άνθρακα στον ενεργειακό μας τομέα μέχρι το 2050 όταν έχουμε στόχο το 27% το 2020 και αυτό ε, είναι ε, λόγω αυξανόμενης ανταγωνιστικότητας. Το 27% θα το επιτύχουμε χωρίς καμία επιπλέον προσπάθεια. Και γι' αυτό θα πρέπει να επιτύχουμε μια συμφωνία ώστε να αυξηθεί αυτός ο στόχος και να συνάδει με ε, το στόχο του 2050. Επιπλέον θα ήθελα να πω ότι ο στόχος που θα θέσουμε θα πρέπει να υπόκειται σε εθνικό επίπεδο και στο εθνικό επίπεδο με δεσμευτικό τρόπο, γιατί το, ε, κάτι άλλο θα ήταν ε, αντιφατικό με τους στόχους. Θέλουμε να έχουμε ανταγωνιστικές ανανεώσιμες ενέργειες και, ε, ηλεκτρική, και, την, να μπορέσει έτσι και η ηλεκτρική αγορά, η αγορά μάλλον ηλεκτρισμού, να συνδεθεί με αυτήν την εξέλιξη. Σημαντικό στοιχείο της οδηγίας είναι ο αρνητικός ε, οικονομικός αντίκτυπος στα project που έχουν ε, ολοκληρωθεί. Είναι πολύ σημαντική αυτή η πτυχή, όμως πρέπει και να ενισχυθεί, να ενισχυθεί η εικόνα της Ευρώπης ως ένα, μια ε, επικράτεια που προσφέρει νομική βεβαιότητα ώστε να γίνουν οι απαραίτητες μεγάλες επενδύσεις που χρειάζονται για να γίνει αυτή η ενεργειακή μετάβαση. Άλλα σημεία κλειδιά της πρότασης είναι να ε, τοποθετηθεί ο καταναλωτής στο επίκεντρο των αποφάσεων ε, για την ε, ενεργειακή απόδοση, δηλαδή η χειραφέτηση του πολίτη, ο συνδυασμός καλύτερων εργαλείων, ε, σύγκριση τιμών και η δυνατότητα να παράγει κανείς και να πουλά την ίδια του την ενέργεια για τον ίδιο αλλά και για τρίτους, αυτό θα σημάνει μια επανάσταση για την αγορά της ενέργειας, γι' αυτό είναι απαραίτητο να προωθηθούν οι ευφυείς λύσεις που έχουν την αυτοκατανάλωση, το ηλεκτρικό αυτοκίνητο, αλλά και την, η διαχείριση όλων αυτών μέσω εφιών δικτύων. Έτσι θα διευκολυνθεί όλη αυτή η διαδικασία που θα ε, χαρακτηρίσει την ε, μελλοντική ενεργειακή αγορά. Να έχουμε δηλαδή ακόμα μια φορά ε, συνοχή, επαναλαμβάνω, για να απελευθερωθεί ο δρόμος ε, και από τεχνικούς, τεχνητούς φραγμούς που τίθεται. Να πω επίσης ότι πρέπει να επιμείνουμε για την ε, συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών ενέργεια στι μεταφορές, γιατί πάνω από το ίμιση των εκπομπών ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλεται ε, στις μεταφορές. Εάν θέλουμε να επιτύχουμε τη μείωση της, χρήση του άνθρακα, θα πρέπει αυτόν τον στόχο να τον θεσπίσουμε. Έχουμε μια Ευρωπαϊκή Ένωση που θέλουμε να προοδεύει και το αποτέλεσμα αυτών των εργασιών θα πρέπει να είναι μια σαφή νομοθεσία που θα είναι κατάλληλη και θα αντιστοιχεί στους στόχους που έχουμε θέσει για την μείωση της χρήσης του άνθρακα. Θέλουμε να βασιστούμε σε μια ενέργεια καθαρή, φθηνότερη και που μάλιστα θα δημιουργήσει και θέσεις απασχόλησης. Γι' αυτό και έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια τεράστια πρόκληση, μια πρόκληση που ταυτόχρονα όμως είναι και μεγάλη ευκαιρία. Thank Σας ευχαριστώ πολύ και τώρα ο σκιώδης εισηγητής για το ΕΛΚ είναι ο κύριος Κέλλη. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς ε, ε, να καλωσορίσω αυτής, αυτές τις προτάσεις ε, για την αναθεώρηση της οδηγίας για την ενέργεια που περιλαμβάνουν διάφορες θετικές, διάφορες θετικά στοιχεία. Να σας πω και ποιες είναι οι βασικές μου σκέψεις από τη μελέτη της πρότασης μέχρι στιγμής. Καταρχάς, με τους στόχους ε, η συζήτηση θα γίνει με την για την στόχο 27% που προτείνεται ως στόχος. Θα πρέπει να θυμίσουμε ότι το Κοινοβούλιο επανειλημμένα έχει εγκρίνει τον υψηλότερο στόχο του 40%. Κάποιοι λένε ότι το 30% είναι πολύ ψηλό ενώ ε, κάποιοι λένε 30% είναι πολύ χαμηλό. Όμως η πλειοψηφία ήταν υπέρ ψηλότερου στόχου στο παρελθόν και γι' αυτό και θα πρέπει να το δούμε όλα αυτά με λεπτομέρειες και να δούμε τελικά ποιος είναι ο πιο ρεαλιστικός στόχο και επίσης θα πρέπει να, μελετή, να δούμε λεπτομέρειες στι μελέτες της ε, Κομισιόν γιατί έχω την εντύπωση ότι το κόστος ορισμένων ανανεώσιμων έχει μειωθεί σε μεγάλο βαθμό Οπότε θα πρέπει να προσπαθήσουμε να ευθυγραμμίσουμε ε, ε την κατάσταση, όμως να μην στείλουμε αρνητικό μήνυμα στις, ε, στη βιομηχανία ανανεώσιμη ενέργεια. Επίσης, να λάβουμε υπόψη ότι το business as usual ε, μπορεί να οδηγήσει στην, στο 27% μείωση μέχρι το 2030 χωρίς καμία επιπλέον προσπάθεια, αν δηλαδή συνεχίσουμε όπως κάνουμε μέχρι τώρα. Ε, ε άρα λοιπόν μήπως πρέπει να αναθεωρηθεί όντως αυτός ο στόχος. Πρέπει περισσότερε ανανεώσιμε να χρησιμοποιηθούν λοιπόν στο ενεργειακό μείγμα, ιδιαίτερα στι περιοχέ τη Υπαίθρου. Είναι σημαντικό η νομοθεσία ως προς αυτό, να προσέξουμε όμως κάποια ζητήματα ώστε να υπάρχει ένα δίκαιο σύστημα ενέργειας οι ε, κοινότητες ουδέτερου, οι ουδέτερες ως προς την ενέργεια θα πρέπει να αναλάβουν το κόστος της διανομής καθώς και της αποθήκευσης, stand-by. Είναι σημαντικό αυτό το κόστος να μην το επιβαρυνθούν όλοι οι καταναλωτές γιατί είναι μικρός ο αριθμός των καταναλωτών που θα ωφεληθούν από αυτές τις ευκαιρίες. Πρέπει να βρούμε λοιπόν μια σωστή ισορροπία. Τώρα, θέρμανση και ψήξη. Επίσης καλώς ορίζω το νέο τμήμα για την θέρμανση και την ψήξη και να πω ότι αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να συζητήσουμε και να εξετάσουμε Τα όσα προτείνει η Κομισιόν ίσως να μην αντικατοπτρίζουν την πολύ γρήγορη πρόοδο που σημειώνεται σε αυτόν τον τομέα. Τέλος να πω ότι πρέπει να δούμε πολύ προσεκτικά ολόκληρο το θέμα των βιοκαυσίμων, γιατί στο παρελθόν έχουμε κάνει λάθος και δεν πρέπει να ξανασφάλουμε. Αυτά για την ώρα, δεν θέλω να μακρηγορήσω άλλο. Ευχαριστώ κύριε Κέλλη. Το λόγο τώρα έχει ο Σκιώδης ε, συγητής του ECR. Ξέρετε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει ένα μερίδιο 27% για τις νόσιμες πηγές ενέργειας για την κατανάλωση ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι το 2030. Το αν θα μείνει αυτό στο 27% ή θα αυξηθεί στο 30% είναι ακόμη υποσυζήτηση. Η συμβολή πάντως κάθε κράτους μέλους θα πρέπει να αποκαθοριστεί, να διασαφινιστεί. Και αυτή τη στιγμή δεν προβλέπονται τομεακοί στόχοι προβλέπ, Οπότε ότι δεν θα χρησιμοποιηθούν νέε ποσοστώσεις όσον αφορά τι ανώσιμε πηγές ενέργειας. Το πρόβλημα είναι βέβαια αυτό το οποίο τίθεται ως απόλυτο ανώτατο όριο για τα βιοκαύσιμα στα μεταφορές από το 7% στο 3,8%. Και εδώ πέρα προβλέπονται οι έμεσες επιπτώσεις της αλλαγής χρήσης της γης θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι υπάρχουν νέα επιχειρηματικά μοντέλα τα οποία προκύπτουν όλο και περισσότερο και τα οποία μπορούν να οδηγήσουν σε πιο οικολογικά βιώσιμα βιοκαύσιμα παντού στην Ευρώπη. Το ερώτημα λοιπόν που τίθεται είναι σε ποιο βαθμό οι Ευρωπαίοι παραγωγοί θα επηρεαστούν από ένα τέτοιο ανώτατο όριο. Επίσης υπάρχουν και κάποιες ανησυχίες από πλευρά των επιστημόνων όσον αφορά τις αρνητικές επιπτώσεις που θα μπορούσε να είχε η χρήση γης και σε άλλες περιοχές, καθότι αυξάνεται η κατανάλωση βιοκαυσίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο εισηγητής μας είπε ότι θα ασχολείται με το ζήτημα του ποσοστού του 27% και θα επιθυμούσε αυτό να περάσει στο 30% βάσει προηγούμενη απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μα είπε επίση ότι συμφωνεί με το ανώτατο όριο που τίθεται για τα συμβατικά βιοκαύσιμα. Επί του παρόντος πρέπει να σας πω ότι είμαι ανοιχτός σε οποιαδήποτε πρότασή σας, δεν έχω καταλήξει κάποια οριστική απόφαση. Πρέπει όμως να πω ότι σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να κάνω υποχωρήσει στο ζήτημα της αρχής επικουρικότητας και ότι θα πρέπει τα κράτη-μέλη πάντα να είναι ελεύθερα να αποφασίζουν ποιο θα είναι το δικό τους ενεργειακό μείγμα. Ο κύριος Φέντερντε τώρα έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Όσον αφορά το στόχο καταρχάς, νομίζω ότι υπάρχει ένα περιθώριο βελτίωσης. Το επ' αυτό και ο εισηγητής. Και από ό,τι κατάλαβα και το ΕΛΚ και το ECR είναι διαλλακτικά ως προς την αύξηση του στόχου αυτού. Νομίζω ότι η Επιτροπή μας η ΙΤΡΕ θα πρέπει να κάνει και μια νέα μελέτη όσον αφορά τις τελευταίες έρευνες που έχουν γίνει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τελευταία αριθμητικά δεδομένα που χρησιμοποιεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι από το 2012, αν δεν κάνω λάθος. Καταλαβαίνετε ότι από το 2012 μέχρι σήμερα δεν έχει ληφθεί υπόψη η εξέλιξη της κοστολόγησης της ενέργειας. Υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη πλέον αλλαγή στις επενδύσεις όσον αφορά τις ανώσιμες πηγές ενέργειας. Γίνονται όλο και περισσότερες επενδύσεις στις ανώσιμες πηγές ενέργειας και το κόστος είναι όλο και πιο χαμηλό. Νομίζω ότι και αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και να επικαιροποιηθούν τα σχετικά δεδομένα. Επίσης το μερίδιο των ανανεώσιμων στη θέρμαση και στην ψήξη και αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη. Υπάρχουν πολλά κράτη-μέλη που έχουν σημαντικό μερίδιο ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στα συστήματα ψήξης και θέρμανσης. Θα πρέπει και αυτό να ληφθεί υπόψη στους συνολικούς στόχους και κατά αυτόν τον τρόπο μπορούμε να φτάσουμε στο 30% μέχρι το 2030. Όσον αφορά τα βιοκαύσιμα, Συμφωνώ με αυτά που είπε ο από το ECR. Νομίζω ότι θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα έχουμε μια γενικότερη μείωση σε εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου χωρίς να κάνουμε επιμέρους διαφοροποιήσεις όσον αφορά τη βιομάζα που προκύπτει από τα δάση. Αυτό αποτελεί εθνική αρμοδιότητα. θα συμπεριληφθεί και αυτό στο ενεργειακό μείγμα των κρατών μελών, θα πρέπει να ακολουθηθεί η εθνική νομοθεσία όσον αφορά τη δασοκομεία και μην ξεχνάμε ότι ε, η κάλυψη από δάση διαφέρει πάρα πολύ από το ένα κράτος μέλος στο άλλο. Υπάρχουν ε, κράτη-μέλη τα οποία καλύπτονται κατά 75 με 80% από δάση, ενώ υπάρχουν άλλα κράτη-μέλη τα οποία ε, έχουν πολύ λιγότερα δάση και δίνουν μάχη αυτή τη στιγμή προκειμένου να καταφέρουν να έχουν μια βιώσιμη δασοκομική πολιτική. Το μερίδιο χρησιμοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έχει μειωθεί τελευταία χρόνια, έχει μειωθεί όμως παράλληλα και το κόστος των πηγών αυτών. Είναι σημαντικό τα επιχειρήματα αυτά να χρησιμοποιηθούν προκειμένου να αυξηθούν οι σχετικές επενδύσεις. Μια έκκληση προς όλους τους συναδέλφους τώρα στην Επιτροπή μας. Έχουμε τεράστια εμείς ευθύνη για το λεγόμενο χειμερινό ενεργειακό πακέτο είναι πάρα πολύ σημαντικό να αντιμετωπίσουμε και την ενδεχόμενη σύγκρουση αρμοδιοτήτων που θα έχουμε μεταξύ κοινοβουλευτικών επιτροπών. Πρέπει να δούμε αν εμείς μπορούμε να αναλάβουμε και το σύστημα ETS ε και το σύνολο της ε, χειμερινής δέσμης μέτρων και να καταφέρουμε ως Επιτροπή Ήτρε να παραμείνουμε σε ηγετική θέση. Ξέρουμε ότι η μάχη θα δοθεί με την Επιτροπή ΕΝΒΗ όσον αφορά τα κριτήρια βιωσιμότητος Νομίζω πάντως ότι θα πρέπει να ορθώσουμε το ανάστημά μας και αν μη τι άλλο να ζητήσουμε συντρέχουσα αρμοδιότητα για όλα τα ζητήματα που άπτονται του χειμερινού πακέτου. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Τούρμες έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, σα ευχαριστώ γιατί από ό,τι φαίνεται έχουμε μια συνένεση αυτή τη στιγμή. Όλοι θεωρούμε ότι το ποσοστό 27% είναι πάρα πολύ χαμηλό. Και είναι πολύ χαμηλό γιατί το κόστο νόσιμων πηγών ενέργεια έχει πέσει. Οι πηγέ αυτές τη ενέργεια ήταν στο παρελθόν ακριβέ. σα δούμε τώρα όμως τι γίνεται με την αιωλική ενέργεια, την ηλιακή ενέργεια, με τις προσφορές που έχουν γίνει στους κλάδους αυτούς το τελευταίο διάστημα και θα συνειδητοποιήσουμε ότι το κόστος έχει μειωθεί πάρα πολύ. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν τα αριθμητικά δεδομένα τη Ευρωπαϊκή Επιτροπής να επικαιροποιηθούν αναλόγως. Αν συνδυάσουμε αυτό με την ευκταία ενεργειακή αποδοτικότητα που θέλουμε να έχουμε, νομίζω ότι μπορούμε πραγματικά να φτάσουμε ακόμα και το 30 και 35% όσον αφορά το μερίδιο χρησιμοποίηση των νεώσιμων πηγών ενέργεια. Πραγματικά δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μα λέει ότι το 50% στην ηλιακή ενέργεια το 2030 είναι το ανώτατο το οποίο μπορούμε να φτάσουμε. Και μετά η, Ευρωπαϊκή Επιτροπή έρθε και μας λέει μας χρησιμοποιούμε την ε, ηλεκτρική θέρμανση, ας χρησιμοποιήσουμε περισσότερο την ηλεκτρική κινητικότητα. Το βρίσκω αυτό αντιφατικό. Καταλαβαίνετε ότι αν δεν προωθήσουμε τη χρησιμοποίηση ηλιακής ενέργειας δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να προωθήσουμε και την ηλεκτρική κινητικότητα. Θα συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε όλο και περισσότερο άνθρακα. Ας μην ξεχνάμε λοιπόν ότι θα πρέπει να συνδυάσουμε τις διαφορετικές πολιτικές μας. Λέμε ότι θέλουμε να προωθήσουμε την ηλεκτρική ε, κινητικό ότι θέλουμε να προωθήσουμε την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων, ότι θέλουμε να έχουμε ηλεκτρική θέρμανση, με αυτό θα πρέπει να συνδυαστεί και με τη χρησιμοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Ακούσαμε διάφορα παραδείγματα. Η Πολωνία, για παράδειγμα, έχει χρησιμοποιήσει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό της επικράτειάς της για την ε, ε, χρησιμοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργεια. Καταλαβαίνουμε όμως ότι πολλές φορές η τιμή της γη, για παράδειγμα, στην Πολωνία είναι πολύ πιο χαμηλή από ό,τι σε άλλες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωση. Και αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι έχουμε 95% χρησιμοποίηση της γης στην Πολωνία, 55% στην Δανία. Το κόστος του κεφαλαίου όμως είναι πολύ πιο ψηλό στην Πολωνία. Αυτό συμβαίνει και με άλλες χώρες. Νομίζω ότι θα πρέπει να επιλύσουμε το πρόβλημα αυτό. Το υψηλότερο κεφαλαιακό κόστος, το οποίο ουσιαστικά λειτουργεί αρνητικά και δεν μας επιτρέπει να χρησιμοποιήσουμε ε, τη γη ακόμα και όταν ε, η τιμή τη είναι πιο χαμηλή. Το ζήτημα τη διακυβέρνηση επίση όσον αφορά τι ανώσιμε πηγέ ενέργεια. Και πάλι εδώ πέρα τα επιχειρήματα προβάλλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι πάρα πολύ αδύναμα. Νομίζω ότι πρέπει να έχουμε εθνικού δεσμευτικού στόχου προκειμένου οι επενδυτέ να έχουν μια κάποια βεβαιότητα και να βοηθήσουμε παράλληλα τα κράτη-μέλη να, να έχουν ωφέλη από τα συστήματα τα οποία χρησιμοποιούμε και στα δίκτυα ενέργειας και στις αγορές ενέργειας. Και στην έκθεση Τσετσίν είχαμε καλύψει και το ζήτημα του κόστους. Θα πρέπει και αυτόν το συνδυάσουμε με τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Να έχουμε ωφέλη κόστους σε διάφορες περιοχές, όπως για παράδειγμα στην Ανατολική Ευρώπη, στην Ιβερική Χερσόνησο, στη Γερμανία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό οι κυβερνήσεις και οι χώρες να καταλάβουν ότι υπάρχουν πάρα πολλές ευκαιρίες εδώ πέρα και ότι ουσιαστικά δεν μιλάμε μόνο για διοικητικό άκθος ή αύξηση του διοικητικού άκθους. Το λόγο έχει η κυρία Λόπες Μπερμέχιο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πραγματικά πραγματικα διερωταμε αν οι υπηρεσίες Ευρωπαϊκής Επιτροπής συνεργάζονται μεταξύ τους, γιατί για το συγκεκριμένο φάκελο από ό,τι φαίνεται ο σχεδιασμός υπολείπεται πάρα πολύ του ευκταίου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε ποιος είναι ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο οποίος από ό,τι φαίνεται εδώ πέρα δεν είναι πάρα πολύ σημαντικός. Νομίζω ότι χρειαζόμαστε μια ενεργειακή μετάβαση η οποία να είναι κοινωνικά δίκαιη, μια καταπολέμηση της ενεργειακής παινίας και ένα εκδημοκρατισμό της παραγωγής και της κατανάλωσης. Και είναι σημαντικό όλοι αυτοί οι παράγοντες να συνδυαστούν μεταξύ τους, να συνδυαστούν τα εθνικά προγράμματα μεταξύ τους, να συνδυαστούν μεταξύ τους οι διάφοροι μηχανισμοί υποστήριξης προκειμένου να προωθήσουμε τις ανανάσιμες πηγές ενέργειας. Δυστυχώς, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πάλι υπολείπεται. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε τα ωφέλη και το κόστος των νόσων πηγών ενέργειας, στην ηλεκτρική ενέργεια, στις μεταφορές, και θα πρέπει βέβαια να προσπιστούμε τα συμφέροντα όλων των εμπλεκόμενων ε, μερών. Δηλαδή να προσπίσουμε και τους μικρούς παραγωγούς. Και είμαι βέβαιη ότι προς αυτήν την κατεύθυνση θα συνεργαστούμε για να φτιάξουμε μια ωραία έκθεση. Ε, Ευχαριστώ Πρόεδρε και εμείς επιβεβαιώνουμε την ευνοϊκή μας θέση υπέρ της παραμονής εθνικών στόχων όσον αφορά τον στόχο της παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας και θα αγωνιστούμε γι' αυτό. Θεωρούμε ότι οι ευρωπαϊκοί στόχοι δεν μπορούν να λειτουργήσουν γιατί το, η δεξιά δεν ξέρετε πήγε αριστερά. Για το νέο deal, ας πούμε, για τον Ευρωπαίο καταναλωτή θα πρέπει να αγωνιστούμε για τα δικαιώματα του καταναλωτή. Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι που η Κομισιόν επέβαλε τις προτάσεις της, όμως θέλω να υπογραμμίσω ότι η συμβολή των καταναλωτών σε, εννοούμε ως πολίτες και παραγωγή ε, θα μπορούσαν να συμβάλλουν σε μεγάλο βαθμό με εντυπωσιακά νούμερα. Αναφέρω μια μελέτη που λέει ότι το 2030 16 ε, εκατομμύρια κόσμος θα μπορούσε να καλύψει μόνος του το 19% της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το 2050 οι μισοί πολίτε θα μπορούσαν να συμμετέχουν δραστήρια ενεργά στην παραγωγή και αποθήκευση ενέργειας αυτόνομα από ανανεώσιμες πηγές, καλύπτοντας το 45% της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Λέγεται πως η Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με τα όσα λέει η Κομισιόν, θα πρέπει να είναι το νούμερο ένα των ανανεώσιμων στον κόσμο. Όμως άλλα στοιχεία από άλλα μέρη του κόσμου δείχνουν ότι αντίθετα υπάρχουν χώρες που προχωρούν πολύ πιο γρήγορα από εμά και ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ενεργειακή Ένωση θα πρέπει να έχει στο επίκεντρό της τον πολίτη και θα δουλέψουμε ώστε αυτό το δύο να μην είναι μόνο συνθήματα, αλλά να αποτελέσουν ρυθμιστικά πλαίσια συνεκτικά, εφαρμόσιμα, ε, ε, έτσι ώστε οι πολίτες πραγματικά να αποτελέσουν τους πρωταγωνιστές της ενεργειακής μετάβασης στην Ευρώπη. Και αυτό χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη όλα τα θετικά ε, πλεονεκτήματα σε περιφερειακό αλλά και σε γεωπολιτικό επίπεδο χάρη στην ανεξαρτησία την ενεργειακή που θα επιτύχουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Ταμπουράνο. Εφτά συνάδελφοι ζητούν για μονόλεπτες παρεμβάσεις. Ο κύριος Κάρινς πρώτος. Ενδιαφέρουσα η συζήτηση. Ένα πρακτικό ζήτημα. Ε, είναι σημαντικός ο φάκελος οι ε, ανακαινήσεις είναι πολύ σημαντικές για πολλά, πολλούς Ένα θέμα πρέπει να σκεφτούμε όμως που έχει να κάνει με τον κανονισμό και το σχεδιασμό της αγοράς. Συχνά όταν έχουμε μέσα έχουμε και διαλύπουσες ή διακοπτόμενες μορφές ενέργειας και εκεί θα χρησιμοποιηθούν τα ορυκτά κάψιμα κάποια στιγμή. Αν θέλουμε να ξεφύγουμε από τις επιδοτήσεις στα ορυκτά θα πρέπει να καταργήσουμε και τις επιδοτήσεις τις ανανεώσιμες γιατί δεν γίνεται το ένα αλλά όχι το άλλο. Δεν θέλουμε να μας τηλεφωνήσει η, ηλεκτρική εταιρεία ότι θα κλείσει το φως. Θα πρέπει να υπάρχει ε, ε, συνέχεια. Δηλαδή, να βρούμε τρόπους να προωθήσουμε τις ανανεώσιμες χωρίς να έχουμε ε, μεγάλη εξάρτηση από επιδοτούμενες μορφές ενέργειας που θα χρησιμοποιούν τα ορυκτά κάψιμα. Ο κύριος Μαρτέν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα επιμείνω σε ένα σημείο το οποίο πραγματικά είναι προβληματικό θεωρώ. Δεν είναι το μόνο πρόβλημα, αλλά είναι αρκετά προβληματικό η πολύ απόλυτη στάση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά την ουδετερότητα, ιδίως για τις διαδικασίες υποβολής προσφορών. Γιατί εδώ πέρα δεν λαμβάνει υπόψη τις τοπικές πτυχές, την καλύτερη τοπική χωροταξία και συγκεκριμένου κλάδους. Να πάρω ένα παράδειγμα. Ας φανταστούμε μια παράκτια περιοχή στην Ευρώπη που θέλει για παράδειγμα να αναπτύξει offshore αιωλικά πάρκα στο μέλλον, με την πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεν θα μπορεί η περιοχή αυτή να πει εκεί θέλω να κάνω επενδύσει και ότι κάνω ένα διαγωνισμό μόνο για να ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια. Ουσιαστικά θα τεθεί σε άμεσο ανταγωνισμό με τι άλλε μορφέ ανανεώσιμων πηγών ενέργεια, με τα φωτοβολταϊκά, τη βιομάζα κτλ. Και αυτή η παράκτεια περιοχή της Ευρώπης θα καταφέρει τελικά να αναπτύξει τον ανανεώσιμο αυτό κλάδο το οποίο θέλει να αναπτύξει. Όπως για παράδειγμα αυτό το οποίο αφορά και τη δική μου την περιφέρεια. Να καταφέρουμε να έχουμε δηλαδή ολικά πάρκα offshore. Αυτό θεωρώ ότι είναι πρόβλημα γιατί ουσιαστικά δεν λαμβάνουμε υπόψη μας την κοινωνία των πολιτών και την τοπική αυτοδιοίκηση η οποία θα πρέπει και αυτή να μπορεί να λαμβάνει κάποιες αποφάσεις. Πολύ καλό να προωθούμε τις νόσιμε πηγές ενέργειας αλλά συνειδητοποιήσουμε ότι όλες οι αρμοδιότητες δεν εξαρτώνται τελικά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο κύριος Κόλιτσεκ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Ο προηγούμενος ομιλητής είπε πολύ σωστά ότι καμιά φορά είναι καλύτερα να χρησιμοποιούμε καμιά φορά ε, ολική, αιωλική ενέργεια ή ε, άλλες φορές Πολλές φορές μπορεί να έχουμε και εφεδρικές πηγές για διακοπτόμενη παραγωγή. Αν χρησιμοποιήσω βιομάζα για ε, φυσικό αέριο και όχι ηλεκτρική ενέργεια άμεσα, μπορεί να έχουμε και ε, την ενέργεια των υδάτων. Ε, μπορεί να υπάρχουν σταθμοί υδροηλεκτρικής ενέργειας και υπάρχουν και μορφές ενέργειας όπως η ολική που θέλει πολύ ή η ηλιακή που χρειάζονται πολύ εφεδρική ενέργεια, υποστήριξη. Η γεωθερμική δεν χρειάζεται. Πώς μπορούμε λοιπόν να έχουμε υποστήριξη ε, ε, αυτών των μορφών ή όταν πρόκειται για μεταφορά ενέργειας. Μιλάμε για το υδρογόνο. Η Ευρωπαϊκή Επιστροπή φαίνεται να μην ενδιαφέρεται γι' αυτό καθόλου. Ενώ το υδρογόνο θα μπορούσε να μας βοηθήσει με τα σκαμπανεβάσματα της κατανάλωσης από τα φωτοβολταϊκά ή τις ανεμογεννήτριες. Υπάρχει λοιπόν δυνατότητα αξιοποίηση και άλλων μορφών. Ευχαριστώ, κύριε Σολίνιο. Τζορίνιο. Σας ευχαριστώ πολύ. Θέλω να χαιρετήσω την εργασία του εισηγητή. Συμμερίζομαι το όραμά του. Η παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές είναι κλειδί για την ενεργειακή μετάβαση και ιδιαίτερα όσον αφορά την ενεργειακή μας επάρκεια και την καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών καθώς και την ενεργειακή ανεξαρτησία μας. Θα προωθηθεί δε με το πρόγραμμα αυτό και η ε, απασχόληση. Όμως πρέπει να είμαστε πιο φιλόδοξοι στους στόχους βασικά ε, για ε, όχι μόνο για τους οικονομικούς λόγους ε, ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι ρυθμίσεις που προβλέπονται από αυτή την οδηγία θα πρέπει να είναι ανάλογες με μια ε, ευφυή ενεργειακή μετάβαση, όπου βασικές γραμμές θα είναι η ένταξη των νεώσιμων πηγών ενέργειας στην αγορά και ο συνδυασμός τους με άλλες μορφές ενέργειας, άλλες πηγές ενέργειας. Για να είναι δίκαιος δε μεταξύ των διαφόρων πηγών θα πρέπει να συνεχίσουμε να στηρίζουμε την έρευνα και την ανάπτυξη σε συστήματα ε, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αλλά και τα συστήματα διανομής. Και επίσης να ηλεκτροδοτηθεί ο τομέας των μεταφορών ε, ε, με ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές. Τέλος, όσον τα συστήματα που υπάρχουν δεν δίνουν πλήρη απάντηση, θα πρέπει να προωθήσουμε τις νέες εξελίξεις, όπως ας πούμε την ενέργεια παράγεται από τα φράγματα, αλλά και την διασύνδεση ανάμεσα στις διάφορες ε, πηγές ενέργειας. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Βέρνε, ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ως σκιώδης παρακολουθώ και την οδηγία αυτή στην Επιτροπή, γιατί οι ανανεώσιμες πηγές είναι πολύ σημαντικές για την αλλαγή στην ενεργειακή αγορά προς ένα όλο και πιο αποκεντρωμένο σύστημα. Ε, η πρόταση της Κομισιόν για την επεξεργασία της ε, οδηγίας για τις ανανεώσιμες έχει πολλά καλά μέτρα. Ε, κάποιες ε, βελτιώσεις όμως χρειάζονται. Πρέπει να είμαστε πιο φιλόδοξοι σε ό,τι αφορά τον καθορισμό των, ε, του μεριδίου των ανανεώσιμων μέχρι το 2030, μετά το 2030. Θα τα συζητήσουμε αυτά. Μπορώ να πω προσωπικά και για την ομάδα μου ότι με το τουλάχιστον 27% χωρίς εθνικά δεσμευτικούς ε, στόχους ε, δεν μπορεί να επιτευχθεί. Δεν είναι αρκετά φιλόδοξο και δεν μας βρίσκει σύμφωνους. Επίσης, θα τονίσω ένα θέμα κυρίως. Στην πρόταση της Κομισιόν ε, επιτρέπονται ε, και στο μέλλον προγράμματα και συστήματα ενίσχυσης. Θα πρέπει όμως να συνάδουν και με την οδηγία για τις επιδοτήσεις. Αλλιώς η διαδικασία θα περιπλακεί πολύ και θα γίνει αδιαφανής. Και τα εθνικά μας υπουργεία θα πρέπει να διαπραγματεύονται επί μήνες με τη Γενική Διεύθυνση ε, για τον ανταγωνισμό για να βρεθούν συμβιβαστικέ λύσεις. Αυτό δεν είναι σωστό. Εμείς θέλουμε ασφάλεια επενδύσεων για τη βιομηχανία και υπάρχουν ε, ήδη εγκεκριμένα συστήματα ενίσχυσης, τα οποία γνωρίζει η Κομισιόν. Θα ήταν πιο αποτελεσματικό λοιπόν να έχουμε έναν κατάλογο κριτηρίων για συστήματα ε, ενίσχυσης και να αποφασίζουμε με την ε, συνήθη ε, νομοθετική διαδικασία. Ευχαριστώ κυρία Βέρνερ. Κυρία Σάντερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να επιμείνω σε δύο δυσκολίες που έχουμε εντοπίσει. Πρώτον, βιοκαύσιμα. Έχουμε τα βιοκαύσιμα πρώτης γενιάς που περνάνε από το 7% στο 3,8% για το 2030 και νομίζω ότι κατά αυτόν τον τρόπο απειλείται ένα ολόκληρο κλάδος και θεωρούμε αυτή τη στιγμή ότι θα προωθηθούν πάρα πολύ και ότι θα αναπτυχθούν πάρα πολύ τα βιοκαύσιμα νέας γενιάς. Το 70% των προτενιών που έχουμε ανάγκη και οι βιοεθανόλοι μπορούν επίσης να βοηθήσουν στη μείωση των απαραίτητων εισαγωγών. Δεύτερον, τεχνολογική ουδετερότητα. Ζήτημα το οποίο δικαλήφθηκε από τους προαλήσαντες. Εδώ δεν υπάρχει σαφήνεια όσον αφορά τη διαδικασία υποβολής προσφορών τεχνολογία οι τοπικές αρχές, η τοπική αυτοδιοίκηση θα πρέπει να μπορούν να ευνοούν τη μία τεχνολογία υπέρ μιας άλλης με βάση της γεωγραφικής τους θέσης, των κλιματικών συνθήκων, της τοπογραφίας και με βάση τον ίδιο του βιομηχανικού κλάδου κλάδους που υφίστανται σε μια περιοχή. Για παράδειγμα, δυνατότητε, γεωθερμίας στην Αλσατία. Χωρί να υπάρχει υποστήριξη για τον κλάδο αυτό, δεν θα καταφέρει ποτέ να αναπτυχθεί και να γίνει όσο ανταγωνιστικέ είναι άλλε τεχνολογίε. Νομίζω ότι οι σημαντικέ συζητήσει θα γίνουν για το ζήτημα αυτό και θα έχουμε τη δυνατότητα να επανέλθουμε στα επιμέρου αυτά ζητήματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Γκρίφιν. Ε, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρέπει να έχουμε νομικό πλαίσιο ενωσιακό ώστε η Ευρώπη να γίνει πρώτη στις ανανεώσιμες πηγές και να υπάρχει ασφάλεια επενδυτών. Η Κομισιόν ε, πρέπει να βελτιώσει την πρότασή της γι' αυτό. Δεν είναι αρκετά φιλόδοξη όπως είπαν αρκετοί συνάδελφοι. Νομίζω ότι πρέπει να έχουμε ε, το δεσμευτικό στόχο 40% και εθνικούς δεσμευτικούς στόχους ούτως ώστε να έχουμε επίτευξη των στόχων στο 2030. Οι κυβερνήσεις ε, θα πρέπει να ενισχυθούν. Πρέπει να τις διαφορές που υπάρχουν να τις λάβουμε υπόψη. Ιδιαίτερα ε, θα πρέπει να βρούμε και τρόπους χρηματοδότησης όπου χρειάζεται. Τώρα, να τελειώσω με κάτι θετικό. Σύμφωνο με τις διατάξεις σχετικά με τις σταθερότητες οικονομικής στήριξης για τα προγράμματα ανανεώσιμων ε, και την αναγνώριση των ενεργειακών κοινοτήτων. Ε, οι πολίτες στο κάτω-κάτω είναι εκείνοι που θα ε, κάνουν την ενεργειακή μετάβαση και νομίζω ότι αυτό που έχει αποδειχθεί είναι ότι πρέπει το πακέτο αυτό να το θεωρήσουμε συνολικά ως πακέτο, ως δέσμη μέτρων. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κουρουμπάσεφ. Κουρουμπάσεφ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να καταλήξουμε σε ένα σύστημα που θα καλύπτουμε τελικά τα πάντα. Ακόμα και ο στόχος αυτός του 27% δεν είναι ρεαλιστικός αν δεν εγκρίνουμε συγκεκριμένους στόχους για κάθε κράτος μέλος. Το ερώτημα αυτό το έθεσα πάρα πολλές φορές στον Επίτροπο Σεφτσοβίτς, αλλά δυστυχώς απάντηση δεν πήρα. Νομίζω λοιπόν ότι το 2014 το Συμβούλιο έλαβε μία απόφαση για το πώς θα καταφέρουμε να διασφαλίσουμε το προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης αν τελικά αγνοήσουμε τη συνεισφορά κάθε κράτους μέλους. Δεύτερον, βλέπουμε εδώ πέρα ότι καταργούνται οι προτιμήσεις. Το δικό μου το κράτος ήταν από τα πρώτα που κάλυψε τους στόχους του στα πλαίσια του προγράμματος με ορίζοντα το 2020. Αν καταργήσουμε όμως τις προτιμησιακές τιμές, ουσιαστικά θα έχουμε 0 μεγαβάτα σε, νέες, σε νέους ε, σταθμούς παραγωγής ενέργειας. Οι νέοι λοιπόν αυτοί κανονισμοί σε καμία περίπτωση θα μας επιτρέψουν να πετύχουμε το στόχο του 27% και σε καμία περίπτωση θα πετύχουμε και πιο φιλόδοξους στόχους βέβαια. Ευχαριστώ. Δεύτερη παρέμβαση του κυρίου Τούρμες. Θα είμαι σύντομος. Η παρατήρηση του κυρίου Καρίνης είναι σημαντική. Ποιο θα είναι το περιβάλλον αγοράς στο μέλλον για όλο το τομέα ηλεκτρικής ενέργειας έχουμε ε, πολύ χαμηλούς στόχους μείωσης του διοξιδίου του άνθρακα. Ε, είχαμε πει ότι θα πρέπει να διπλασιάσουμε την αποθηκευτική ικανότητα στην Ευρώπη. Ε, αυτό είχε γίνει το 2002-2004 και είχαμε τότε μεγάλα σκαμπανεβάσματα. Τώρα είναι χαμηλό το ε, διοξίδιο του άνθρακα. Και το spread είναι ε, μικρό. Η ευελιξία που έχουμε στο σύστημα ε, δεν αντιμετωπίζεται με τόσο χαμηλή τιμή διοξιδίου του άνθρακα. Ε, διότι αν είναι τόσο χαμηλή η τιμή για το διοξίδιο του άνθρακα θα υπάρχει χαμηλή διάχυση. Μπορεί λοιπόν να, να πρέπει να δώσουμε ε, κίνητρα ούτω ώστε να λειτουργήσουν εναλλακτικέ μορφές. Οι αναλύσεις της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού είναι χρήσιμες εδώ. Η Γενική Διεύθυνση ε, δέχεται ότι μπορεί να γίνει ένα χρηματοδότηση στην αγορά για ορισμένες ε, ε, νέες μορφές. Thank you. Are Ευχαριστώ. Άλλες παρεμβάσεις δεν υπάρχουν. Τότε να δώσουμε το λόγο στην Κομισιόν. Η κυρία Αμπρό Μαρκές για τρία λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Πρέπει να πω ότι η Κομισιόν χαίρεται που βλέπει το ενδιαφέρον που δημιούργησε η πρωτοβουλία αυτή, όπως φάνηκε σήμερα. Η αναθεώρηση της οδηγίας θέλει να δημιουργήσει ένα θετικό πλαίσιο για τα κράτη-μέλη ώστε να ανανεώσουν το ενεργειακό δυναμικό τους και να φτάσουν στο 27% ανανεώσιμων μέχρι το 2030. Όπως ε, είπε και ο κ. Μπλάνκο και άλλοι, πράγματι είναι σημαντική νομοθετική πρόταση για να ε, κάνει την Ευρωπαϊκή Ένωση πρώτη στις ανανεώσιμες και οι καταναλωτές να, μείνουν να είναι στο επίκεντρο. Το Κοινοβούλιο κατά το παρελθόν ήταν υπέρ του τουλάχιστον 30%. Με βάση τη, πολλά μοντέλα που καταρτήσαμε ε, με το 27% έχουμε, ε, βλέπουμε ότι το 2030 θα μπορέσουμε να επιτύχουμε και το στόχο του άνθρακα, χρήσης του άνθρακα. Ε, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το 2014, τον Οκτώβριο, είχε δεχτεί την πρόταση της Κομισιόν. Οι, κύριοι Φέντερλε, και Τούρμες ε, ανέφεραν την εκτίμηση επιπτώσεων που πολλές φορές επεκρίθη διότι ε, χρησιμοποίησε μη ρεαλιστικές τιμές ε, και κόστη για κάποιες ανανεώσιμες. Διευκρινίζομαι ότι τα ποσά αυτά ήταν ενδεικτικά. Παραδείγματα. Ε, χρησιμοποιεί η Κομισιόν το μοντέλο Primes που δίνει ένα συνολικό σύστημα μοντέλων και οι υποθέσεις κόστου στηρίζονται στα πιο ενημερωμένα δεδομένα. Θα είμαστε ευτυχείς να ε, βελτιώσουμε και να δώσουμε και πληροφορίες περισσότερες στο μέλλον. Ε, Επίση, ε, έχουμε και άλλες φιλοδοξίες, όχι μόνο στόχους. Έχουμε υπόψη μας να καλύψουμε τον τομέα της ενέργειας, ειδικότερα στου διάφορους τομείς, θέρμανση, ψήξη κλπ. Να βελτιώσουμε τις επενδύσεις του ανανεώσιμες. Ε, υπάρχουν και διατάξεις στην ε, οδηγία για το, τη διακυβέρνηση, την ενεργειακή απόδοση κλπ. Ε, θα ήθελα να απαντήσω και σε ορισμένα σχόλια που έγιναν και αυτό το θέμα. Καταρχήν, να προωθούμε πιο σύντονη και οργανωμένη προσέγγιση για προγράμματα στήριξη των κρατών μελών που θα στηρίζονται περισσότερο στην αγορά, ώστε να ελαχιστοποιούνται οι στρεβλώσει αγορά και να χρησιμοποιούνται οι ανανεώσιμε πηγέ όσο πιο αποτελεσματικά σε σχέση με το κόστο γίνεται σε όλη την Ευρώπη, όπω είπε και ο κ. Κάρεν. Ε, ενθαρρύνομαι ε, αναδιόμενες ε, τεχνολογίες. Θέλουμε να προωθήσουμε την καινοτομία. Ε, Επίση ε, προβλέπουμε αλλαγές με αναδρομική ισχύ. Θέλουμε να προωθήσουμε την διαφάνεια στους κανονισμούς, κανονιστική ασφάλεια που χρειάζεται για να μειώσουμε το κεφαλαιοχικό κόστος, όπως είπε και ο κύριος Τούρμες. Επίσης βλέπουμε και στην ψήξη και στη θέρμανση το δυναμικό των ανανεώσιμων, 50% της κατανάλωσης. Επίσης, όπως είπα, πρέπει να φτάσουμε το 25% με τρόπο ε, αποτελεσματικό σε σχέση με το κόστος. Θέλουμε αύξηση κατά 1% των ανανεώσιμων για κάθε κράτος μέλος και να έχουμε άνοιγμα προς τους ε, παραγωγούς που εφοδιάζουν με ανανεώσιμες πηγές. Επίσης, ε, θέλουμε κίνητρα ε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο στο σκέλος της ε, προσφοράς ανανεώσιμων. Θέλουμε επίσης να έχουμε και ειδική εντολή για προηγμένα βιοκαύσιμα. Επίσης δίνουμε τη δυνατότητα στους καταναλωτές και απαντώ εδώ στον κύριο Ταμπουράνο ατομικά ή με οργανωμένο τρόπο σε κοινότητες να ε, παραγάγουν ενέργεια και να την αποθηκεύουν χωρίς ε, ε, δυσανάλογα βάρη. Και οι καταναλωτές που συμβάλλουν στο κόστος, στο ναι, σύστημα, σε ένα σύστημα ενέργειας, θα έχουν ανάλογη μείωση των τελών. Επίσης, Υπάρχει διαδικασία απλουστευμένη για μικρής κλίμακας έργα και κατοπορισμένε συνθήκες για την ε, ε, ανακαίνιση υφισταμένων ε, ε, μονάδων. Ε, εδώ έχουμε μεγάλη μείωση παραγωγής εκπομπών θερμοκηπίου σε σχέση με τα ορυκτά καύσιμα χωρίς απώλεια βιοδιαφοροποίησης ε, υπ' αυτή την έννοια να αναφέρω ότι η πρόταση ε, ευθυγραμμίζεται απόλυτα με την εθνική αρμοδιότητα των κρατών μελών. Η πρόταση αυτή έχει σαφείς διασυνδέσεις με άλλες νομοθετικές προτάσεις στο, στη δέσμη καθαρής ενέργειας, αυτή για τη διακυβέρνηση και την πρωτοβουλία για το σχεδιασμό της αγοράς. Ο στόχος λοιπόν που, όλοι, που έχουμε κοινό είναι να έχουμε συνοχή, ε, μέτρα συνεπή για την περίοδο μετά το 2020 που θα οδηγήσουν στην αναγκαία ενεργειακή μετάβαση στην Ένωση. Η Κομισιόν προσβλέπει σε συνεχείς και επικοδομητικές συζητήσεις για την αναθεώρηση της οδηγίας με το Κοινοβούλιο η φιλοδοξία είναι ε, για να ε, υλοποιήσουμε τις φιλοδοξίες μας ε, που θα οδηγήσουν σε μεγαλύτερη απασχόληση και βεβαίως θα ωφεληθούμε και από το μειούμενο κόστος της τεχνολογίας. Ευχαριστώ. Και τώρα για να ολοκληρώσουμε, κυρία Μπλάνκο Λόπες. Σας ευχαριστώ όλους για τους σκέψεις που διατυπώσατε και για τις προτάσεις και θέλω να κάνω έτσι ενθερμό κάποιες παρατηρήσεις. Ε, μετά από αυτή την ενδιαφέρουσα συζήτηση. Ήδη ε, με την έκθεση Λόπις Βερμέχο πολλά από τα πράγματα που έχουμε πει ε, τα έχουμε ξαναπεί. Γι' αυτό και πιστεύω ότι όταν θέτουμε ένα γενικό στόχο του 27% οικομεσιών, το θέτει αυτό το στόχο, αυτό δεν συνάδει ούτε με τους στόχους που έχουμε ορίσει για το 2050, αλλά ούτε και λαμβάνουν υπόψη τη μείωση τους, ε, του κόστους ε, της ενέργειας που προέρχεται από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που έχουν οριμάσει. Άρα λοιπόν το 27% είναι μάλιστα και κακό μήνυμα γιατί εκτός που δεν είναι φιλόδοξο δείχνει ότι δεν ε, Έχουμε λάβει υπόψη πως η τεχνολογία έχει προχωρήσει και είναι σε αρκετά όριμο στάδιο που να επιτρέπει την παραγωγή σε πολύ πιο χαμηλό κόστος και άρα ε, και επιτρέπει την επίτευξη πιο, πολύ πιο φιλόδοξων στόχων από αυτούς που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και επίσης ε, δεν προσφέρει, και εδώ θέλω να πω το εξή, δεν προσφέρει ένα σαφές μήνυμα ε, με το, τις απαραίτητες επενδύσεις. Έχουμε μιλήσει επί μακρόν για το τι είναι απαραίτητο στο να εγγυηθούμε την ε, ε, νομική βεβαιότητα γιατί ξέρουμε τι έγινε σε κάποιες χώρες ε, με αναδρομικές διατάξεις κτλ. Λοιπόν, γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό το να το θέσουμε και αυτό. Εάν θέλουμε πραγματικά να προσελκύσουμε επενδύσεις, εάν θέλουμε οι επενδύσεις αυτές να γίνουν με βιώσιμο και μόνιμο τρόπο, εάν δεν τεθούν δεσμευτικοί στόχοι σε επίπεδο των χωρών, δεν ε, θα γίνουν ε, επενδύσεις που να ρισκάρουν εφόσον η ε, δεσμευτική στόχη δεν είναι σαφής. Να κάνουμε λοιπόν μια παραπάνω προσπάθεια ώστε να εξασφαλίσουμε την νομική βεβαιότητα δεν έχει νόημα εάν δεν θέσουμε εθνικούς στόχους. Αυτό πρέπει να το λύσουμε το πρόβλημα, γιατί διαφορετικά δεν θα προχωρήσουμε αρκετά. Ε, επίσης, ε, θα πρέπει να γίνει και συζήτηση για τα βιοκαύσιμα πρώτης και δεύτερης γενιάς. Ε, να συζητήσουμε την οδηγία που στόχο έχει μια, ένα είδος ισορροπίας. Δεν ξέρω αν είναι επαρκές, ε, αλλά πάντως πρέπει να σκεφτούμε ότι ο τομέας των μεταφορών είναι αυτός ο οποίος μολύνει περισσότερο, ρηπαίνει περισσότερο και άρα πρέπει και να γίνει μια παραπάνω προσπάθεια. Ο στόχος του 10% για τη τρέχουσα περίοδο δεν είναι επαρκής. Πρέπει να γίνει μια παραπάνω προσπάθεια σε αυτόν τον τομέα που είναι αυτός που ρηπαίνει περισσότερο και δεν πρέπει να το ξεχνάμε τη στιγμή που μιλάμε για αυτή την οδηγία. Και να μην ε, ξεχνάμε και τα όσα είπαμε για την ε, παραγωγή και κατανάλωση, αυτοκατανάλωση. Πρέπει να το λάβουμε αυτό υπόψη γιατί είναι καινούριο αυτό. Γιατί επιπλέον ε, χειραφετεί τον πολίτη κάθετο καταναλωτή συμβάλλει στην μείωση της χρήσης του άνθρακα. Ε, πρέπει λοιπόν να μην το ξεχνάμε και να αναζητήσουμε τα μέτρα που θεσπίζουν ισορροπία αλλά που μας επιτρέπουν να στείλουμε σαφή μηνύματα και να θεσπίσουμε φιλόδοξους στόχους ε, καθώς και να μην οπισθοδρομήσουμε. Κατά τη γνώμη μου λοιπόν, όπω είπα, η μη δεσμευτική στόχη για τα κράτη είναι ένα βήμα πίσω. Θα πρέπει να συνεχίσουμε να το συζητάμε και εγώ ήδη ε, ευχαριστώ για όλε σας τι συμβολέ και είμαι βέβαιο ότι θα καταφέρουμε να κάνουμε καλή έκθεση. Σα ευχαριστώ πολύ συνάδελφοι για τι συμβολέ σα και για την πειθαρχία σα να σας ενημερώσω ότι το σχέδιο έκθεση αναμένεται ε, ε, για τις 29 και 30 ε, Μαΐου. Απόψε η συνεδρίαση της Επιτροπής μας επίσης να σας θυμίσω ότι θα γίνει στην PHS 5 Β1, δηλαδή στον 5ο όροφο αίθουσα Β1 και θα ξεκινήσουμε στις 15.45, 4 παρατέταρτο και όχι στις 3 και θα προεδρεύσει η πρώτη μας αντιπρόεδρος η κυρία Τόγια.